Buongiorno. Καλημέρα. Buongiorno. Καλημέρα παρακαλώ. Καθίστε. Ευχαριστώ. Να σας υπενθυμίσω πως η αίθουσα 3C050 είναι συνδεδεμένη με την αίθουσα της Ολομέλειας για να επιτραπεί στους βουλευτές που δεν μπορούν να καθίσουν στην Ολομέλεια να μπορέσουν να συμμετάσχουν στην διαδικασία με τους κανόνες της απόστασης. Όσοι είναι στον κατάλογο των ομιλητών παρακαλώ να έρθουν να καθίσουν εδώ στο ημικύκλιο όπου θα βρουν στο έδρανό τους ε, με ένα χαρτί με το όνομά τους. Όσοι δεν είναι στον κατάλογο παρακαλώ να ακολουθήσουν τους κλητήρες τα υπόλοιπα διαθέσιμα έδρανα. Σας ενημερώνω πως υπάρχει παρουσιολόγιο και στις δύο αίθουσες και υπενθυμίζω επίσης πως η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική. Όσοι θέλουν να παρέμβουν χωρίς μάσκα μπορούν να το κάνουν μόνο για την διάρκεια της ομιλίας τους. Άρχεται λοιπόν η συνεδρίαση η οποία είχε διακοπεί στις 15 Μαΐου 2020. Τα πρακτικά τι 13, 13 Τρίτης, ε, Τετάρτης και Πέμπτης σας έχουν μοιραστεί. Υπάρχουν παρατηρησει Όχι. Οπότε εγκρίνονται. Κάποιες ανακοινωσει Η ομάδα ECR με ενημέρωσε για μια απόφαση αλλαγή όσον αφορά τον διορισμό σε μια αντιπροσωπεία. Η απόφαση αυτή θα περιληφθεί στα πρακτικά της σημερινή συνεδρίασης. Να ενημερώσω την αίθουσα πω σύμφωνα με το άρθρο 79 του κανονισμού υπέγραψα μας με τον πρόεδρο του Συμβουλίου 7 νομοθετικές πράξεις οι οποίες είχαν εγκριθεί με βάση την τακτική νομοθετική διαδικασία. Οι τίτλοι θα δημοσιευτούν στα πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης. Περνάμε τώρα στην διάταξη των εργασιών το σχέδιο μερίσια διάταξη που έχει εγκρίνει στις 19 Μαΐου η διάσκεψη των Προέδρων σύμφωνα με το άρθρο 177 σας έχει μοιραστεί. Δεν έχει ζητηθεί κάποια άλλαγη της ημερήσιας διάταξης. Οπότε εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη και η διάταξη των εργασιών. Περνάμε τώρα στην συζήτηση, δήλωση της Κομισιόν και του Συμβουλίου για το θέμα Ευρωπαϊκό Σχέδιο Οικονομικής Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να υπενθυμίσω στους βουλευτές πως ε, δεν προβλέπεται διαδικασία και ούτε μπλε κάρτα. Να χαιρετήσω την ε, πρόεδρο, την κυρία Φόντερ Λάιν, που είναι παρούσα εδώ, μαζί με όλους τους επιτρόπους. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Τον λόγο έχει εξ ονόματος του Συμβουλίου η Υπουργός κυρία Μπρινιέτς. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να πω λίγα λόγια για το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάκαμψης που θα υποβάλει σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι κάτι πολύ καινούριο ακόμη και οι αντιπροσωπείες τώρα άρχισαν να το εξετάζουν. Ω εκ τούτου, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είμαι ακόμη σε θέση να επισέλθω στην ουσία των προτάσεων τη δέσμη μέτρων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα έχουμε και άλλε ευκαιρίε για κάτι τέτοιο. Θα ήθελα προ το παρόν να υπενθυμίσω πώ η Προεδρία σκοπεύει να προχωρήσει από εδώ και πέρα. Καταρχήν, να ξεκινήσω με κάποιε προσδοκίε. Στα τέλη Απριλίου, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων αποφάσισαν να συσταθεί ένα ταμείο ανάκαμψη και το έκριναν ω εκτάκτο ανάγκη. Και προσδοκούν ότι θα είναι δεόντως ε, πρικοδοτημένο ε, που και θα στηρίξει τους τομείς και τις περιφέρειες που έχουν πληγεί περισσότερο για να ανταπεξέλθουν σε αυτή την πρωτοφανή κρίση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε ως καθήκον να εξετάσει τις ε, άμεσες ανάγκες και να υποβάλει κατεπηγόντως μια πρόταση που θα ανταπεξέλθει στο ύψος των προκλήσεών μας. Περιμένω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσδιορίσει τη σχέση του νέου ταμείου με το πολιετέ δημονομικό πλαίσιο, που με βάση τη γνώμη των ηγετών θα πρέπει να προσαρμοστεί στην τρέχουσα κρίση και τι συνέπειε και τα επακολουθά τη. Αναλαμβάνοντα αυτό το καθήκον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προετοίμασε ένα περιεκτικό πακέτο των οριζόντιων προτάσεων που θα μα υποβάλει σήμερα. Οι πολιτικέ οδηγίε ήταν σαφεί. Οι αντιπροσωπείε θα εξετάσουν το πακέτο υπό το φω αυτό των προσδοκιών και θα ξεκινήσουν από τώρα την ανάλυση των λεπτομεριών. Σε ό,τι αφορά την διοργάνωση των εργασιών, το, η λέξη κλειδί είναι ε, κατεπίγουσα διαδικασία υπάρχει έκτακτη ανάγκη. Και μάλιστα και τον περασμένο μήνα οι ηγέτε εξέφρασαν την επιθυμία να καταλήξουν συμφωνία το συντομότερο δυνατό. Ο χρόνο τρέχει. Θα πρέπει να προχωρήσουμε και να αποφασίσουμε το συντομότερο δυνατό. Το απαιτούν οι οικονομίε μα και το περιμένουν οι πολίτε μα. Είναι ευθύνη τη Προεδρία λοιπόν να προωθήσει τι εργασίε ε, πάρα αυτά και χωρί χρονοτριβή υπό το φω τη πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και μάλιστα οι Υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν. Ε, ένα, συνολικό πακέτο ανάκαμψης με έναν προσαρμοσμένο πιδελταπή και μηχανισμό ανάκαμψης. Επιπλέον, θέσαμε στην ημερήσια διάταξη του Κορεπέρ για πρώτη προκαταρκτική συζήτηση αμέσω μετά την παρουσίαση του πακέτου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήδη σήμερα μία πρώτη συνάντηση των μόνιμων αντιπροσώπων. Θα χρειαστεί φυσικά και τεχνική προεργασία για να προετοιμαστεί η ανάλυση των προτάσεων πριν καταλήξουν σε ουσιαστική ε, συζήτηση οι ηγέτε. Γι' αυτό και το Συμβούλιο και με αυτοπρόσωπη παρουσίαση και με τη βοήθεια της τεχνολογίας θα εγγύψει σε αυτό. Περιμένουμε φυσικά ε, και θα λάβουμε υπόψη τις αποφάσεις του Ευρω... της του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και λάβαμε υπόψη και το ψήφισμά σας ε, για το νέο πιδελταπή, τους ιδίους πόρους και το σχέδιο ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είχα αναφέρει και τότε, η συνεχή συνεργασία μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα της διαδικασίας και σε οριζόντιο επίπεδο αλλά και σε τομιακό επίπεδο. Επί τη ευκαιρία θα ήθελα να σα υπενθυμίσω ότι πέραν τη συμφωνία για το ΠΙΔΕΛΤΑΠΗ έχουμε και δεκάδε άλλε διαπραγματεύσει που αφορούν προγράμματα που μετατρέπουν την ευρωπαϊκή υποστήριξη σε έμπρακτη εφαρμογή. Και φυσικά ο χρόνο πιέζει. Θα πρέπει και στο τομεακό επίπεδο να σημειώσουμε όση περισσότερη πρόοδο γίνεται. Έχουμε ελάχιστο χρόνο και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε στου μελλοντικού δικαιούχου των προγραμμάτων, τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, του φοιτητέ, την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλου, τη συνέχιση. Σήμερα περισσότερο από ποτέ χρειάζονται τη στήριξή μα για να δρομολογηθούν και να εφαρμοστούν τα προγράμματά του. Έτσι θα βοηθήσουμε την ανάκαμψη της οικονομίας μας, των περιφερειών μας και των πολιτών μας και προσβλέπουμε σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις προσδοκίες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Υπουργέ. Τον λόγο τώρα έχει η κυρία Φόντερ Λάιεν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η Ευρώπη είναι μια ιστορία γενεών και κάθε ευρωπαϊκή γενεά έχει τη δική της ιστορία. Για τη γενιά που ίδρυσε την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ιστορία έκανε λόγο για τη δημιουργία βιώσιμης ειρήνης, ειρήνης διαρκείας, όταν υπήρχε μόνο οδύνη, πόνος, καταστροφή. Για την επόμενη γενιά, ο στόχος ήταν η ευημερία και η ελευθερία να εδρεωθούν, να παγιωθούν. Επιλέξαμε την ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς και ένα κοινό νόμισμα. Εν συνεχεία, το θέμα ήταν η ευρωπαϊκή οικογένεια να ενωθεί, οι αδελφοί να βγουν και να ενταχθούν ε, στην οικογένειά μας, να τους υποδεχθούμε εδώ στο επίκεντρο, στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλες αυτές οι γενιές και όλες αυτές οι ιστορικές επιτυχίες οικοδομήθηκαν και εμπνεύστηκαν ε, από τους πολεότερους για τους νεότερους. Ο στόχος ήταν να προχωρήσει κανείς από μόνος του ή από κοινού όλοι μαζί, με, με ένα κοινό όραμα, με μια φιλοδοξία κοινή και προς την ίδια κατεύθυνση. Σε αυτές τις αποφασιστικές ε, στιγμές και ώρες αποφασίσαμε πάντοτε να κάνουμε ένα βήμα προς τα εμπρός όλοι μαζί, ένα άλμα όλοι μαζί προς τα εμπρός. Χρειάζεται μια πιο θαραλέα Ευρώπη γιατί έτσι θα είμαστε και πιο ασφαλείς. Και αυτό μας, μας έδωσε τη δυνατότητα να οικοδομήσουμε αυτή την ένωση της ειρήνης και της ευημερία που δεν έχει προηγούμενο ε, και ούτε και κάτι αντίστοιχο έχουμε δει σε κάποιο άλλο μέρος του κόσμου μέχρι τώρα. Αγαπητοί ευρωβουλευτές. Σήμερα είμαστε αντιμέτωποι με μια ακόμη καθοριστική χρονική στιγμή. Αυτό που ξεκίνησε με έναν ιό τόσο μικρό στο μάτι που κανείς δεν μπορεί να τον δει ουσιαστικά, έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη οικονομική κρίση που κανείς δεν μπορεί να κάνει ότι δεν τη βλέπει. Το μοναδικό μας μοντέλο που ε, δημιουργήθηκε μέσα σε αυτά τα 70 χρόνια που πέρασαν έχει δεχθεί μια πρόκληση άνευ προηγουμένου στην ιστορία της κοινής ευρωπαϊκής ιστορίας έχουμε προβλήματα, ε, αντιμφισβητούνται πράγματα που θεωρούσαμε δεδομένα. Πρέπει να ανακάμψει όμως η ευρωπαϊκή αγορά. Πρέπει να έχουμε ξανά ένα ισότιμο πεδίο για όλους και να αποκαταστήσουμε πλήρως τις ελευθερίες. Η κρίση έχει πάρα πολύ σημαντικές εξωτερικές και δευτερογενείς επιπτώσεις παντού. Και τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί να τα φτιάξει από μόνη τη, να τα διορθώσει από μόνη τη κάποια χώρα χωρίς τη συνδρομή των άλλων. γιατί μια χώρα μπορεί να είναι προμηθευτής ε, ή ε, αποδέκτης ε, μιας άλλης και θέλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι αν είναι αποδυναμωμένη η οικονομία μιας χώρας αποδυναμώνεται η οικονομία και στις άλλες χώρες. Επομένως είναι κάτι που μας ξεπερνά και δεν έχει να κάνει με, με κάτι που αφορά τον καθένα από εμά, έχει να κάνει με την Ευρώπη συνολικά. Όλα τα κράτη-μέλη ε, πλήττονται. Οι ανισότητες ε, βλέπουμε να ε, οξύνονται. Το χάσμα να διευρύνεται. Έχουμε ζητήματα που άπτονται της, του κράτους δικαίου και της αλληλεγγύης και πρέπει να τα εξορροπήσουμε όλα αυτά. Και έχουμε πάλι την ίδια διτή επιλογή ή θα προχωρήσει ο καθένας από μόνος του αφήνοντας χώρες, περιοχές και ανθρώπους πίσω και να δεχθούμε την Ευρώπη όπου κάποιοι έχουν και κάποιοι δεν έχουν ή θα προχωρήσουμε μαζί αυτό το μονοπάτι, θα κάνουμε μαζί το άλμα και θα κάνουμε ένα γερό βήμα προς τα εμπρός για το λαό μας, ε, για τους λαούς μας και για τις επόμενες γενναίες. Για μένα είναι μια απλή επιλογή. Εγώ θέλω να κάνουμε ένα γενναίο βήμα όλοι μαζί προς τα εμπρός. Η Ευρώπη βρίσκεται σε μια μοναδική θέση. Μπορεί να επενδύσει στη συλλογική ανάκαμψη, στο κοινό μέλλον. Στην Ένωσή μας οι άνθρωποι, επιχειρήσεις, εταιρείε εξαρτώνται ένας από τον άλλο, βασίζονται ένας στον άλλο. Στην Ένωση μας η συνοχή, η σύγκληση, οι επενδύσεις είναι ένα κοινό αγαθό, έχουν ωφέλη για όλους. Και γνωρίζουμε στην Ένωση ότι τα πιο θαραλέα, τα πιο γενναία μέτρα είναι τα πιο ασφαλή, πραγματικά τα πιο ασφαλή για το μέλλον. Και αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα καταθέτει ένα νέο ε, μέσο ε, για την ανάκαμψη που λέγεται Next Generation EU. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση της επόμενης γενιάς με 750 δις ευρώ τα οποία έρχονται να προσθεθούν στο ανανεωμένο ε, μακροπρόθεσμο δημοσιονομικό σχέδιο του 1,23 εκατομμυρίου με το Next Generation και με το ΠΔΠ έχουμε 1,85 δισεκατομμύρια στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή. Και αυτό μαζί ε, στα 540 δις που είναι ένα δίκτυο ασφαλείας που έχουν ήδη συμφωνήσει Κοινοβούλιο και Συμβούλιο. Και θεωρούμε ότι με, με αυτή την προσπάθεια θα έχουμε πολλές δυνατότητες να πετύχουμε την ανάκαψη με 2,43 ευρώ. Τρέψατε μου αγαπητοί ευρωβουλευτές να σας εξηγήσω το πώς θα λειτουργήσει αυτό το νέο εργαλείο Next Generation EU. Τα χρήματα θα τα συγκεντρώσουμε έροντας ε, τα ανώτατες οροφές ε, στους ίδιους πόρους. Ε, θα μπορεί δηλαδή η Ένωση να δανείζεται στις αγορές λόγω της προνομιακής της θέσης με πολύ ευνοϊκούς όρους. Αυτό είναι μια αναγκαιότητα, είναι κάτι αναγκαίο γιατί βρισκόμαστε σε μια έκτακτη κατάσταση, βρισκόμαστε σε εποχή κρίσης. Το Next Generation EU θα επενδύσει στην αποκατάσταση του κοινωνικού ιστού, στην προστασία της ενιαίας εσωτερικής αγοράς θα βοηθήσει να υπάρξει ο σκέλος των προπολογισμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και θα πρέπει να πατήσουμε το fast forward και να προχωρήσουμε με πιο ταχύ βήμα ε, προς ε, μια πράσινη οικονομία, ένα νέο μέλλον, γιατί αυτό είναι το μέλλον της ε, νέας γενιάς, next generation μιας γενιά συνδεδεμένης ε, που ε, θέλει να αναλάβει την υποχρέωση για την προστασία του πλανήτη. Θέλουμε επίση να προστατεύσουμε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το κράτος δικαίου να ε, είναι πιο υπεύθυνε και να λογοδοτούν οι κυβερνήσεις ότι αντιμετωπίζουν πράγματι την κλιματική αλλαγή, ότι σώζουν τη φύση ιδεολογία ε, υπέρ της Ευρώπης, πίστη ε, στην Ένωση ότι μπορεί να αγωνιστεί και να πετύχει περισσότερα. Άρα δεν χρειάζεται μόνο αλληλεγγύη για να ξεπεράσουμε σήμερα την κρίση. Θέλω να προτείνω και ε, ένα σύμφωνο για τη νέα γενναία, για το μέλλον. Γιατί ναι, πράγματι η κρίση αυτή σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν επενδύσεις σε άνευ προηγουμένου κλίμακα. Σήμερα αυτό. Και θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε όμως με έναν τρόπο ώστε η επόμενη γενιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορεί να δρέψει τους καρπούς αυτής της σημερινής προσπάθειας. Οι επενδύσεις αυτές δεν θα διατηρήσουν μόνο τα εξαιρετικά επιτεύγματα των τελευταίων 70 ετών. Θα εξασφαλίσουν ακόμη το ότι είναι κλιματικά ουδέτερη ένωση, το ότι είναι ψηφιακή, κοινωνική και ισχυρό παγκόσμιο πρωταγωνιστή και σήμερα και στο μέλλον. Και για να γίνει αυτό πραγματικότητα, επόμενη γενιά, ε, το Next Generation EU, το μεγάλο μέρος του θα το διαθέσει σε κοινέ προτεραιότητες μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Αξιότιμοι βουλευτές, ε, θέλω πάντοτε ε, να γνωρίζετε ότι θέλω να εξασφαλίσω ότι θα έχετε ως Κοινοβούλιο πάντοτε λόγο σε αυτές τις εξελίξεις κρίσμες. Η πρόταση ε, για να επενδύσουμε μέσω προγραμμάτων σε αυτούς τους στόχους ακριβώς εκεί αποσκοπεί. Το Next Generation EU ουσιαστικά θα αποκαταστήσει την ενιαία αυτή αγορά που γεννά καινοτομία, ευκαιρίες, ευημερία. Όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να επενδύουν, να επενδύσουν σε τεχνολογίες ε, που θα πυροδοτήσουν εκ νέου την ανάκαψη, με καινοτομία, με καθαρές βιομηχανίες. Το Next Generation EU ενισχύει και την Πράσινη Συμφωνία και τον Οριζοντα Ευρώπη θα ε, επενδύσουμε από το 5G σε μέτρα για την ε, ανακαίνιση κτηρίων, ε, θα προωθήσουμε την κλιματική ουδετερότητα, αλλά ταυτόχρονα θα φροντίσουμε να μην μείνει κανείς πίσω. Το Next Generation EU, επομένως, θα πολλαπλασιάσει ουσιαστικά τη χρηματοδότηση του Ταμείου Δικής Μετάβασης. Και πάντα στο ίδιο πνεύμα, κανένα κράτος μέλος δεν θα πρέπει να κληθεί να, επιστρέ... να επιλέξει αν θα γυρίσει πίσω στην κρίση ή θα επενδύσει στους ανθρώπους. Γι' αυτό λοιπόν ε, θα αυξηθεί ε, η πρικοδότηση του Εράσμου και η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων επίση θα ενισχυθεί μέσω του Next Generation. Για να έχει ο κόσμο δεξιότητε, ε, δουλειέ, θα πρέπει να μπορεί να προσαρμοστεί στον ταχύω μεταβαλλόμενο κόσμο, ιδίω η νέα γενιά. Το Next Generation EU θα βοηθήσει επίσης τις υγιείς αυτές επιχειρήσεις που κάνανε ε, τα σωστά βήματα, που πήραν ε, τις σωστές αποφάσεις ε, επενδύοντας τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά τώρα βρίσκονται σε κίνδυνο γιατί οι ανταγωνιστές από άλλα κράτη-μέλη έχουν καλύτερη πρόσβαση στους δημόσιους ιδιωτικούς πόρους θα επενδύσουμε σε βασικές τεχνολογίες και βιομηχανίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να είναι πιο ανθεκτικές οι βασικές αλυσίδες ε, εφοδιασμού ώστε η Ευρώπη να παραμείνει στην αιχμή, ε, στην προτεραιότητα σε ό,τι αφορά παραδείγματο χάρη την γεωργία ακριβία, ε, την πράσινη μηχανική ή την τεχνητή νοημοσύνη. Και το Next Generation EU θα φροντίσει να είναι πιο ανθεκτικά γενικώ τα συστήματα, να μπορούν να αντέξουν μελλοντικέ κρίσει. Αυτέ οι επενδύσει θα είναι ένα νέο κοινό ευρωπαϊκό αγαθό. Θα δείξουν την πραγματική, την απτή αξία της συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση του ανήκεν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι κάτι το οποίο θα το κάνουμε όλοι κτήμα μας, όλοι θα το ιδιοποιηθούμε. 750 δις για το Next Generation EU θα συλλεγούν. Τα 500 δις ε, εξ αυτών θα είναι σε επιχορηγήσεις, θα τεθούν σε επιχορηγήσεις και τα 250 σε δάνεια προς τα κράτη-μέλη. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, να είμαι σαφής. Αυτά, αυτές οι επιδοτήσεις είναι μια κοινή επένδυση στο μέλλον μας. Δεν έχουν δε μια σχέση με τα χρέη των κρατών του παρελθόντος. Οι επιδοτήσει περνάνε από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και υπάρχει μια συγκεκριμένη κλίδα κατανομής. Πηγαίνουν ξεκάθαρα ως επενδύσεις στις ευρωπαϊκές μας προτεραιότητες, στην ενίσχυση της εσωτερική αγοράς, στην ψηφιοποίηση, στο ευρωπαϊκό Green Deal, στην ανθεκτικότητα και άλλα. Ο ευρωπαϊκό προπολογισμό πάντα, πάντα ήταν επιδοτήσεις. Δεν είναι κάτι το νέο επιδοτήσεις για στοχευμένες επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις, για περισσότερη συνοχή επιδοτήσεις για να υπάρξει σύγκληση του επίπεδου ζωής στην Ευρώπη. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η ζωντανή απόδειξη για το ότι αυτό λειτουργεί. Έτσι αυξήθηκε η ανταγωνιστικότητα και το επίπεδο ζωής κάθε κράτους μέλους. Κάθε κράτου μέλους. Η επένδυση αυτή μέσω του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού έχει αποδώσει για όλους το πολλαπλάσιο. Και το ίδιο ισχύει και για το Next Generation EU. Επενδύουμε μαζί στο μέλλον της Ευρώπης και έχουμε βεβαίως την γνωστή κλίδα και επιπλέον η Κομισιόν θα προτείνει μία σειρά νέων ίδιων πόρων που θα μπορούσαν παραδείγματο χάρη να είναι η επέκταση του εμπορίου εκπομπών ή έναν φόρο διοξιδίου του άνθρακα στα σύνορα το οποίο θα αφορά τα φτηνότερα προϊόντα που εισάγονται και βλάπτουν το περιβάλλον για να υπάρξει μια συνεισφορά στην κοινή μας ευημερία. Και εδώ πέρα θέλω την στήριξή σας. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, τώρα είναι η στιγμή να λάβουμε τις κατάλληλες αποφάσεις. Αυτοί οι οποίοι σήμερα δεν θέλουν να γίνουν θαραλέες επενδύσεις σε αυτούς λέω ότι θα πληρώσουμε αύριο το κόστος του να μην κάνουμε τίποτα. Πρέπει να θέσουμε τις βάσεις για το κοινό μας μέλλον. Και ταυτόχρονα να έχουμε την δυνατότητα να αντιδράσουμε ξεκάθαρα σε μια κρίση άνευ προηγουμένου. Οπότε πρέπει να ξεπεράσουμε τις προκαταλήψεις μας, να ανακαλύψουμε και πάλι την δύναμη που προκύπτει από αυτή τη μεγάλη ιδέα μιας κοινή Ευρώπης. Είναι μεγάλη η πρόκληση, αλλά εξίσου μεγάλη είναι η ευκαιρία για την Ευρώπη και η ευθύνη μας να κάνουμε το σωστό σε αυτή την κατάσταση. Τώρα μπορούμε να θέσουμε τις βάσεις για μια ένωση η οποία θα είναι κλιματικά ουδέτερη, ψηφιακή, εύρωστη και θα έχει καλύτερη αντιμετώπιση των κοινωνικών ζητημάτων. Για 70 χρόνια οι ίδρυτες έκαναν πριν από 70 χρόνια, έκαναν τα πρώτα βήματα για μια ένωση της ειρήνης και της ευημερίας. Σήμερα είναι η στιγμή να προσθέσουμε το κεφάλαιο της δικής μας γενιάς και να κάνουμε ένα παραπέρα θαραλέο βήμα σε μια ένωση της αηφορίας. Το οφείλουμε στις επόμενες γενιές. Ζήτω η Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Ε, Σας ε, ευχαριστώ ε, κυρία Πρόεδρε. Πριν να ακούσουμε τους πρόεδρους των πολιτικών ομάδων θα ήθελα η βουλευτές ε, από τους οποίους ζητήθηκε να φύγουν από τα έδρανα για λόγους ασφαλείας να το σεβαστούν. Ε, συνάδελφε, κύριε, στο 34, σας το έχουν πει ήδη δύο φορές. Παρακαλώ να σεβαστείτε. Ο κύριος Μάνφρετ Βέμπερ έχει το λόγο. Ε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, Αγαπητοί συνάδελφοι, η αλληλεγγύη έχει επανέλθει, η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, το πνεύμα του Ρομπέρ Σουμάν. Πριν από λίγε εβδομάδε έκαιγαν ευρωπαϊκέ σημαίε στην Ιταλία. Εκατομμύρια άνθρωποι ανησυχούν ακόμα και φοβούνται για το μέλλον του, για τι οικογένειε του για τι δουλειέ του. Η Ευρώπη σήμερα δίνει μια δυνατή απάντηση. Δεν είστε μόνοι. Μαζί θα ανταποκριθούμε, θα δώσουμε την κατάλληλη απάντηση με μια αλληλεγγύη. Ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αγαπητοί συνάδελφοι, κάποιοι αποκάλυψαν την τωρινή στιγμή μια στιγμή Χάμιλτον. Δεν μου αρέσει βέβαια ως πολιτικός του Έλκα. Εγώ δεν θέλω να βασίζεται η Ευρώπη στα χρέη, αλλά έχοντας όλα αυτά κατά νου, την κρίση, τη μεγαλύτερη κρίση από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τώρα έχει φτάσει η στιγμή να επενδύσουμε, να δώσουμε μια νέα όθηση στην οικονομία μας. Αλλά το βασικό ερώτημα για εμάς δεν είναι πρώτα απ' όλα πόσο μεγάλη θα είναι η επένδυση, πόσα λεφτά θα ξοδέψουμε. Δεν είναι αυτό το βασικότερο. Το πρώτο ερώτημα είναι πού θα πάνε τα λεφτά, γιατί χρειάζονται. Και έχουμε τώρα μια πρόταση η οποία εγγυάται ότι δεν θα δώσουμε νέα λεφτά για τα παλιά προβλήματα. Θα δώσουμε νέα χρήματα για νέες ιδέε για ένα νέο μέλλον για αυτή την Ήπειρο. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο είναι κρίσιμο για εμάς στην συζήτηση είναι οι δημοκρατικέ διαδικασίες και ευχαριστώ την πρόεδρο της Κομισιόν ε, για την δήλωσή τη. Τώρα πρέπει να πάμε στο Συμβούλιο και να ξεκαθαρίσει με το Συμβούλιο ότι η αρχή πώ δεν θα ξοδεύονται λεφτά στο ευρωπαϊκό επίπεδο ε, χωρίς τον έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να υλοποιηθεί. Επίσης, πρέπει να πείσουμε 27 κράτη-μέλη, κοινοβούλια, για να στηριχθεί αυτή η ιδέα. Και είναι περίεργο να βλέπουμε ότι στο ΕΛΚ έχουμε μία κυβέρνηση, έχουμε δύο σοσιαλιστικές κυβερνήσεις, μία φιλελεύθερη κυβέρνηση στον Αντιάκομα και οι πράσινοι είναι μέρος του προβλήματος, γιατί στην Αυστρία κυβερνούν Οπότε χαίρομαι που βλέπω ότι όλοι μας έχουμε την ίδια πρόκληση να πείσουμε τους άλλους να στηρίξουν την γενική αυτή ιδέα. Και για τις ε, τέσσερις χώρες ε, που είναι εναντίον από το εξή. Πρώτα απ' όλα, οι δικές σας οι δεν μπορούν να είναι ε, επιτυχείς χωρίς την ενιαία αγορά, οπότε είναι προς το συμφέρον σας να καταστήσετε επιτυχία ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δεύτερο επιχείρημα, βλέπουμε μια ανακατανομή της παγκόσμιας οικονομικής ισχύω και δεν θα ήθελα να κερδίσει η Κίνα και να χάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και 2008-2010 ήδη αντιμετωπίσαμε το φαινόμενο μιας χαμένης γενιάς. Η Ευρώπη δεν μπορεί να δεχτεί άλλη μια χαμένη γενιά αυτή τη φορά. Γι' αυτό νομίζω πως έχουμε καλά επιχειρήματα για να σας πείσουμε. Για εμάς η αλληλεγγύη πάει χέρι με χέρι με την ευθύνη. Είναι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος για μας το ΕΛΚ. Και έχοντας αυτό κατά νου, σας λέω το εξής ότι όταν πηγαίνουμε σε αγορές και δανειζόμαστε λεφτά, πρέπει να είμαστε σαφείς να έχουμε ξεκάθαρες ιδέες για το πώς θα αποπληρώσουμε. Και να πούμε ότι στο επόμενο πι δελτα πι, όταν θα γίνει η συζήτηση, είχε ξεκινήσει βεβαίω ήδη το Μάρτιο και προσπαθούσε το Συμβούλιο να βρει κάποια συμφωνία. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη φορά θα είναι τόσο εύκολα. Γι' αυτό εμείς ω ΕΛΚ πρέπει να είμαστε ειλικρινεί, σαφείς και αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε ίδιους πόρου για να πληρώσουμε το χρέος που έχουμε τώρα. Ο μεγάλος νικητής τη κρίση είναι οι ψηφιακοί γίγαντες, γι' αυτό νομίζω ότι είναι δίκαιο να του ζητήσουμε να πληρώσουν κομμάτι του χρέου που δημιουργούμε. Και ένα άλλο τμήμα αυτή τη ευθύνη αλληλεγγύη. είναι η εθνική πτυχή. Μπορείτε να το πείτε εξάμεινο, μπορείτε να το πείτε ανάγκη εσωτερικών μεταρρυθμίσεων. Νομίζω ότι είναι δίκαιο αν ζητάμε από τον γείτονα να μας βοηθήσει με αλληλεγγύη να κάνει και ο καθένα αυτό που το αναλογεί για να είναι πιο προετοιμασμένο για το μέλλον. Και σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο χρειαζόμαστε μεταρρυθμίσει. Υπάρχουν και άλλε αρχέ που είναι σημαντικέ. Το κράτο δικαίου. Εμεί ε, το υποστηρίζουμε. Νομίζω έχουμε μια καλή συμβαστική πρόταση. Το πρόγραμμα επίσης έχει αναβαθμιστεί ε, για την υγεία. Ένα σημαντικό μήνυμα σε καιρούς κορονοϊού. Θα γίνουν και άλλες συζητήσεις και βέβαια έχουμε και τη γεωργία και τη συνοχή. Οπότε το σχέδιο πηγαίνει σε καλή κατεύθυνση. Είναι μια σημαντική στιγμή για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ΕΛΚ σε γενικές γραμμές θα στηρίξει τις ιδέες της Κομισιόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, η κυρία Γκαρσία Ένα μήνα μετά την έγκριση του ψηφίσματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, είστε εδώ και μας παρουσιάζετε το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάκαμψης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι φιλόδοξο το σχέδιό σας, είναι φιλοευρωπαϊκό το σχέδιό σας και είναι ένα σχέδιο που ακολουθεί τις διεκδικήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και σας ευχαριστώ που δώσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το ρόλο που το αξίζει. Μας βάλατε σε ισότιμη θέση με το Συμβούλιο σε ό,τι αφορά το σχέδιο ανάκαμψης ε, και τη συζήτηση για τους ίδιους πόρους και το ΠΔΠ. Επίσης, το σχέδιο σας περιλαμβάνει την έκδοση ομολόγων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Χρέος. Ε, έτσι επιτρέπεται στα κράτη-μέλη να χρηματοδοτηθούν με δίκαιο τρόπο για να αντιμετωπίσουν αυτή την κρίση. Είναι προφανές ότι κάτι έχει αλλάξει. Κάποιε προτάσει που συμπεριλάβατε στο σχέδιό σα και που ε, ήδη τι υποστήριξαν κάποιε κυβερνήσει θα ήταν αδιανόητε πριν από μερικού μήνε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πολλές εθνικές κυβερνήσεις έχουν συνειδητοποιήσει το μείζον διακύβευμα που είναι το μέλλον και η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μιλούμε μόνο για αλληλεγγύη αλλά για την επιβίωση του ευρώ και της ενιαίας αγοράς, της εσωτερικής αγοράς. Και φυσικά σε τελική ανάλυση μιλούμε και για την επιβίωση του ευρωπαϊκού σχεδίου. Γιατί μερικοί ίσως δεν έχουν αντιληφθεί ακόμη ότι εδώ δεν είμαστε για να κάνουμε αγορά τουλάχιστον η δική μου πολιτική ομάδα δεν ενδιαφέρεται για την αγορά, αλλά για τη δημιουργία τη συγκρότηση μια πολιτική ένωση. Μερικοί στο Συμβούλιο μιλάνε σαν να μην συνέβη τίποτα. Σαν οι τελευταίοι μήνε ε, ε, να μην ε, μα έφεραν την τεράστια κρίση, σαν να μην είχαν χάσει τη ζωή του 160.000 άνθρωποι στην Ευρώπη, σαν να μην είχε τεθεί σε κίνδυνο η εργασία πάνω από 60 εκατομμυρίων ε, Ευρωπαίων, σαν να μην γνωρίζαμε ότι η κρίση αυτή θα προκαλέσει μια τεράστια ύφεση και ότι το ΑΕΠ της Ευρωζώνης θα συρρικνωθεί κατά 8% φέτος. Αν όλα αυτά λοιπόν δεν μας εξωθήσουν να αναλάβουμε δράση, τότε τι περιμένουν μερικοί. Είναι η στιγμή της αλήθειας. Θα πρέπει να ανοίξουμε τα χαρτιά μας. Θα πρέπει, θέλουμε να συνεχίσουμε να δημιουργούμε μια πολιτική ένωση, γιατί αυτό ξεπερνάει την αλληλεγγύη. Και επίσης θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι σε αυτόν τον ταραγμένο κόσμο, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να εργαστούμε για να προασπίσουμε το ευρωπαϊκό σχέδιο. Η κρίση COVID-19 είναι συμμετρική κρίση με ασύμετρα αποτελέσματα. Και το θεμελιώδη ζήτημα εδώ είναι, πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διορθώσει τις ασυμμετρίες. Γιατί δεν έχει νόημα να ασχολούμαστε και να επεξεργαζόμαστε ένα κοινό σχέδιο και μετά να αφήνουμε μερικέ επιχειρήσει να βοηθούν τι, ε, μερικέ χώρε να βοηθούν τι επιχειρήσει του, ενώ άλλε χώρε επειδή δεν έχουν πόρου αφήνουν τι επιχειρήσει του να χρεοκοπήσουν. Ή θα γλιτώσουμε όλοι ή δεν θα γλιτώσει κανένα. Αν κάποιοι στο Συμβούλιο δεν πιστεύουν στι ευρωπαϊκέ λύσει και στη σύγκληση, τότε δεν θα πρέπει τουλάχιστον να παρεμποδίζουν την πορεία των άλλων που είναι υπέρ τη Ευρώπη. Α είμαστε ειλικρινεί. Το πρόβλημα δεν είναι τα χρήματα, τα περισσότερα κονδύλια. Το πρόβλημα είναι να προχωρήσουμε στην Ευρώπη. Γι' αυτό το Συμβούλιο θα πρέπει να τροποποιήσει τη διαδικασία για την, για την έγκριση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου και να περάσει από την ομοφωνία στην ενισχυμένη πλειοψηφία. Γιατί είναι άδικο 23 φιλοευρωπαϊκέ χώρε να γίνουν όμοιροι εχμάλωτοι των τεσσάρων που προτιμούν τι εθνικέ μεταρρυθμίσει πέραν της έλλειψη αλληλεγγύης, κάτι τέτοιο είναι μια κοντόφθαλμη συμπεριφορά ομοιοπική. Γιατί αρκεί να ρίξει μια ματιά κανείς γύρω του για να αντιληφθεί ότι η πολυμέρεια βρίσκεται σε κίνδυνο και χρειαζόμαστε μια παγκόσμια διακυβέρνηση. Θα πρέπει επίση να ενισχύσουμε τον κοινωνικό πυλώνα, να προστατεύσουμε αυτού που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Και χαίρομαι που συμπεριλάβατε και την εγγύηση για τα παιδιά. Είναι καθήκον μας να δείξουμε αλληλεγγύη προς τις επερχόμενες γενιές και να επενδύσουμε στις σημαντικές πολιτικές για το μέλλον. Με, μετασχηματισμός ψηφιακός, φιλοπεριβαλλοντικός, γιατί δεν μπορούμε να, βάζουμε, να, να διακυβεύουμε το μέλλον του περιβάλλοντος και να επιβαρύνουμε τις επερχόμενες γενιές με τεράστια χρέη. Συμφωνώ με την πρόταση για την αλλαγή του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Θα πρέπει να ξεπεράσουμε την λογική της ε, δημοσιονομικής εξυγίανσης. Θα πρέπει να επενδύσουμε στη βιωσιμότητα και την κοινωνική και την περιβαλλοντική. Αυτό το μέλλον που θέλουμε να σφυριλατήσουμε από κοινού θα πρέπει να στηρίζεται και στην ε, υποστήριξη του κράτου δικαίου. Θα πρέπει να υπομισθούμε τι ευθύνε μα, αγαπητοί συνάδελφοι. Κυρία Φοντερ Λάιν, είδατε ότι εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχετε συμμάχου και έχουμε ένα σχέδιο που θέλουμε να θέσουμε ε, στη, στους Ευρωπαίους πολίτες. Ελπίζω να πείσουμε και το Συμβούλιο. Να, είσ, να δείξετε πυγμή, να είστε φιλόδοξοι και θα μας βρείτε στο πλευρό σας. Γιατί αυτό οφείλουμε στις επόμενες γενιές των Ευρωπαίων. Ευχαριστώ. Κύριε Τσόλο, έχετε τον λόγο. Ο κύριο Τσόλο έχει τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Πραγματικά αλλάζει τα δεδομένα αυτή η κρίση που αντιμετωπίζουμε. Είναι κάτι άνευ προηγουμένου στην ιστορία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μέγεθο, οι διαστάσει τη κρίση, οι εξαιρετικέ προκλήσει τη απαιτούν και μία ανάλογη και γρήγορη αντίδραση. Εναλλακτική άλλη δεν υπάρχει και η λύση είναι η μαζική ε, σε επενδύσει στην οικονομία, αλλιώ δεχόμαστε ότι θα πληγούμε και ακόμα πιο σφοδρά. Πρόκειται για μια δέσμη μέτρων για όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό πρέπει να είναι σαφέ. Όλα τα κράτη-μέλη χρειάζονται αυτή τη δέσμη μέτρων, αυτό το πακέτο ανεξαρτήτως το πόσο βαριά επλήγησαν από αυτήν την υγειονομική και οικονομική κρίση, διότι εδώ διακυβεύεται το μέλλον της εσωτερικής αγοράς. Αν αποτύχει η εσωτερική αγορά, όλοι οι πολίτες, όλες οι επιχειρήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης θα υποφέρουν. Η λύση της Προέδρου Φοντρελάιεν να δανειστεί δηλαδή από τις αγορές ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Χρήματα είναι μια λύση που πρέπει να πούμε ότι είναι ε, αξιοσημείωτη, αξιοπρόσεκτη. Ευρωπαϊκή λύση για ευρωπαϊκό πρόβλημα. Ε, είναι θετικό αυτό. Επίση, αποφεύγεται μια σημαντική δυσκολία που αντιμετωπίσαμε στην τελευταία αυτή κρίση. Δημιουργία δηλαδή περισσότερου χρέου για κάποια κράτη-μέλη από τη στιγμή που χρειάζονται χρήματα τα οποία θα τα ε, διοχετεύσουν άμεσα στι οικονομίε του. Οι αποφάσει που λαμβάνουμε τώρα ε, θα διαμορφώσουν το μέλλον μα τα επόμενα 20-30 χρόνια και το ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον. Γιατί ο στόχο μα είναι να κινήσει εκ νέου, να δρομολογηθεί εκ νέου η ανάπτυξη και η οικονομία. Δουλεύουμε για τι επόμενε γενναίε. Ακριβώ γι' αυτό αυτό το πακέτο ανάκαμψη ε, και ε, το νέο ΠΔΕΛΤΑΠΗ θα πρέπει να ε, σκέφτονται να είναι στραμμένα προ το μέλλον και να μην βασίζονται σε πεπαλαιωμένε αντιλήψει. Θέλουμε να δημιουργήσουμε νέε θέσει εργασία, να επενδύσουμε μάλλον να ε, ενισχύσουμε τι επενδύσει ε, σε έργα τα οποία έχουν πραγματική οικονομική προσθέμενη αξία και θα οικοδομήσουμε έτσι μια κυρίαρχη ανθεκτική οικονομία. ή αλληλεγγύη. η αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη είναι σημείο κλειδί. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τι εδαφικέ ανισότητες, ε, το εδαφικό χάσμα. Αυτό είναι ένα πρόσφορο έδαφο για την Ένωση. Αν δεν το πετύχουμε θα σπείρουμε σπόρου μελλοντική διχόνοια. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Τρίτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά δεν είναι ε, μια μηχανή που κόβει χρήμα. Είναι μια λέγκια ε, διαδικασία με κοινέ αρχέ, κοινέ αξίε, κοινό όραμα για το μέλλον. Η ομάδα μας, το Renew Europe, θα στηρίξει το ΠΔΠ μόνο εκεί που το κράτος δικαίου και ο σεβασμός των ευρωπαϊκών αξιών είναι προϋπόθεση για να λάβει μια χώρα ευρωπαϊκά κονδύλια. Δεν θέλουμε να τιμωρήσουμε τους απλούς πολίτες, αλλά τους πολιτικούς οι οποίοι δεν τηρούν τους κανόνες. Σε τέταρτον, Σίγουρα έχουμε πολλά διδάγματα να αντιλήσουμε από την κρίση αυτή <clears throat> για να βελτιώσουμε, να μεταρρυθμίσουμε τομεί που εκεί πρέπει να είναι πιο παρούσα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν η διάσκεψη για το μέλλον τη Ευρώπη, για το κοινό μα μέλλον, πρέπει κάποια στιγμή να ξεκινήσει. Θα είναι δύσκολο και μακρύ το μονοπάτι προς την ανάκαμψη και οι αποφάσεις που λαμβάνουμε τώρα θα επηρεάσουν τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων, όπως και το μέλλον της, οικονομικής, της ε, αγοράς της Ένωσης, ε, της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Πρέπει να είμαστε ενωμένοι και πρέπει να αγωνιστούμε ως ένας. Μία γροθιά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τσιόλος, λέει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. Μόιτεν, παρακαλώ, εξ ονόματος ομάδας ID, κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε της ε, Κομισιόν. Η κυρία Μέρκελ τα είπε ξεκάθαρα ούτε ευρωομόλογα ούτε κορονοομόλογα. Και τώρα, τώρα μιλάτε για ένα ταμείο οικοδόμησης 500 δισεκατομμυρίων. Το τεράστιο αυτό ποσό το οποίο θα χρηματοδοτηθεί πρώτα με επιστώσεις ε, και μετά από τους φορολογούμενους. Χωρί κάποια νομική βάση βεβαίω, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή δεν έχει ίδιου πόρου. Κάτι το οποίο φαίνεται δεν σα ενοχλεί. Και τώρα έρχεστε εδώ πέρα, κυρία Πρόεδρε τη Κομισιόν, και απαιτείτε η τρέλα αυτή να μην αρκεί, θέλετε άλλα 250 δισεκατομμύρια στην διάθεσή σας. Αυτό είναι, σας το λέω, ξεκάθαρα τρέλα. Γιατί το τίμημα αυτό θα το πληρώσουν οι πολίτες πάρα πολύ ακριβά. Τα λεφτά αυτά δεν είναι δικά σας, είναι των πολιτών. Αυτό το οποίο κάνετε είναι τελείως ανέθινο. Είναι οικονομικά βουντού είναι χαρακτήρι και οικονομικής και νομισματικής πολιτικής. Βεβαίω ο κόσμος έχει αυτή τη στιγμή άλλε ανησυχίε που τον απασχολούν. Και αυτό εκμεταλλεύεστε εσείς με τις παράλογες απαιτήσει, τις οποίες ονομάζεται μάλιστα τελείως υποκριτικά αλληλεγγύη. Απευθύνω έκκληση στις κυβερνήσεις Αυστρίας, Δανίας, Ολλανδίας και Σουηδίας να σταματήσουν να αρνηθούν αυτήν την τρέλα. Σας ευχαριστώ. Κυρία Κέλλερ, έχετε τον λόγο. Thank Σας ευχαριστώ. Όντως, ε, περνάμε μια βαθύτατη κρίση στην Ευρώπη και θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Είναι μια στιγμή μεγάλης ευθύνης Σκεφτόμαστε λοιπόν να συνεργαστούμε και να εξέλθουμε από κοινό από αυτή την κρίση. Και στο Κοινοβούλιο με μεγάλη πλειοψηφία δείξαμε τη σωστή άγουσα. Με ένα ταμείο ανάκαμψης, με ένα ισχυρό προϋπολογισμό και μια πράσινη συμφωνία που θα βοηθήσει την οικονομία, ενώ ταυτόχρονα θα αντιμετωπίσει την κλιματική κρίση και την κρίση βιοπικιλότητας, που δεν πάει πουθενά. Γιατί η πράσινη παντού στην Ευρώπη είναι υπέρ αυτής της ε, προσέγγισης και Αγαπητέ Βέμπερ, είναι πραγματικά φθηνό να κρύβεστε πίσω από του πράσινου όταν υπάρχει μεγάλη και λαϊκή υποστήριξη και στην Αυστρία υπέρ των θέσεων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ίσως ο καλός σας φίλος στη Βιέννη δημιουργεί πρόβλημα. Αλλά χαίρομαι που δείξετε κι εσείς μια προθυμία να το μεταπίσετε. Και εκεί μπορούμε να συνεργαστούμε για να προσπαθήσουμε από κοινού να μεταπίσουμε τις κυβερνήσεις, ε, τα κόμματα παντού υπέρ αυτής της κατεύθυνσης, γιατί αυτό θα πρέπει να κάνουμε τώρα. Πάντως πιστεύω ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ένα μεγάλο βήμα προόδου και χαιρετίζουμε το ότι επικεντρώνεστε στις επιχορηγήσεις, ώστε να μην μείνει πίσω στην κρίση κανένα καμία χώρα. Ίσως μπορεί ε, μακροπρόθεσμα να μην ε, αρκέσουν αυτά τα κονδύλια. Πάντως σε καμία περίπτωση θα πρέπει να μειώσουμε τις φιλοδοξίες μας στο ΠΔΠ, γιατί θα πρέπει να έχουμε υπόψη και το μέλλον. Αναφέρθηκαν πολλοί συνάδελφοι σε προποθέσει σε όρου που θα πρέπει να συνδυαστούν με το Ταμείο. Αλλά παρακαλώ, α μην επαναλάβουμε τα κολοσσία λάθη του παρελθόντο και να αναγκάσουμε τι χώρε ε, σε μια πολιτική λιτότητα ή τυφλή πολιτική οικονομική υπέρ τη αγορά που δεν θα οδηγήσει πουθενά. Θα πρέπει να επενδύσουμε σωστά τα κονδύλια αυτά σε μακροπρόθεσμα προγράμματα που θα δημιουργήσουν θέσει απασχόληση και θα σώσουν τον ένα και μοναδικό πλανήτη που έχουμε. Επίσης, μέσω και μέσω μακροπρόθεσμα και το ΠΙΔΕΛΤΑΠΗ και το Ταμείο Ανάκαμψη θα πρέπει να δώσουν κίνητρα για την κοινωνική ε, μετατροπή τη κοινωνίας και για την ε, αποκατάσταση της ισότητας των φύλων. Επίσης θα πρέπει να έχουμε ελάχιστους κοινού αγώνες, ε, κανόνες όπως του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας. Δεν μπορεί μία χώρα μόνη της να αντιμετωπίσει την κρίση, γιατί όλες οι χώρες έχουμε αποφεληθεί από την ε, εσωτερική αγορά, την ελεύθερη διακίνηση και μάλιστα μερικές χώρες αποφελήθηκαν και από τους υπερβολικά χαλαρούς φορολογικούς κανόνες. Θα πρέπει λοιπόν να εντείνουμε τις δράσεις μας, όπως έκαναν και οι ιδρυτές πατέρες, ο Σούμαν πριν από 70 χρόνια. Και το Κοινοβούλιο έχει δείξει ετοιμότητα να αναλάβει και να διαδραματίσει το ρόλο του. Ελπίζω να μας ακολουθήσουν και τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τέρ Όφερφελντ, εξ του ECR, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, έχω εντυπωσιαστεί πολύ από το πώς οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μας μπόρεσαν να αντιδράσουν με τρόπο ευέλικτο και δυναμικό στην κρίση. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Τα μέτρα μας πρέπει να είναι αποτελεσματικά. Βεβαίω όταν μιλάμε για δάνεια και επιδοτήσει, πρέπει να υπάρχουν κάποιοι όροι που συνδέονται με αυτά. Και βεβαίω ε, πρέπει να ληφθούν και μέτρα τα οποία δεν κοστίζουν άμεσα λεφτά. Η ενίσχυση της ε, εσωτερικής αγοράς απολύτω αναγκαία και πρέπει να φροντίσουμε να προστατεύσουμε τις επιχειρήσεις μας. Ε, διεθνείς όμιλοι συγκεντρώνουν μυθικά ποσά χωρίς να έχουν τις καλύτερες των ε, προθέσεων. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει ένας μηχανισμός προστασίας. Βεβαίω ε, το θέμα είναι του που θα βρεθούν τα λεφτά, αλλά και πρέπει να δούμε και το θέμα της ε, χρηματοδότησης, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται και αποταμιεύουν δεν μπορεί να ματώνουν από αυτήν την υπόθεση. Επιπλέον πρέπει να αντιληφθούμε ότι υπάρχουν κάποια όρια στον τρόπο και στην ένταση με την οποία χρησιμοποιούμε τις δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας γιατί συχνά δημιουργείται η εντύπωση πως πρόκειται για α, χρήμα χωρίς τέλος. Ενώ αυτό δεν ε, ισχύει. Θα πρέπει επίσης ε, να δούμε την ε, συζήτηση που αφορά την συμβολή των γιγάντων του διαδικτύου οι οποίοι συμβάλλουν πάρα πολύ λίγο και θα πρέπει να συμβάλλουν αυτό που τους αναλογεί. Αυτό θα πρέπει να γίνει αποτελεσματικά. Και οπωσδήποτε ε, θα πρέπει τώρα να αναλάβει και η Ευρώπη τον ρόλο που της αναλογεί. Σας ευχαριστώ. Ομπρί, έχετε τον λόγο. Κύριε Ομπρή, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Φοντερ είναι εδώ και μήνες σας είχαμε προειδοποιήσει ότι δεν είναι παρένθεση αυτή η κρίση φαίνεται να ε, έχει τις ρίζες της ε, στις πολιτικές που εξάντλησαν ε, το σύστημα υγείας των χωρών, κατέστρεψαν το μηχανικό ιστό και την προστασία, την κοινωνική. Μας μιλάτε για τις γενές και τη νέα γενιά. Εγώ είμαι ακριβώ μέλος αυτής της γενιάς η οποία υπέστη την καταστροφική δράση των νεοφιλελεύθερων πολιτικών που δημιούργησαν ανισότητες και κατέστρεψαν τον πλανήτη. Αυτό το σχέδιο ανάκαμψης που μας παρουσιάζεται σήμερα θα έπρεπε να συνιστά τομή, ξεκάθαρη τομή με τις πολιτικές του παρελθόντος αλλά δυστυχώς ε, ε, μένει στη μέση ε, και μια μιλάτε για τη λιτότητα ότι είναι πίσω μας πια και στην αρχή της κρίσης είχαν πάψει να ισχύουν κάποια τέτοια μέτρα τώρα όμως από, το, από την πίσω πόρτα επανέρχεται με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο με την επιβολή όρων και προϋποθέσεων προς τα κράτη-μέλη για να επανέλθει κοινωνική ισορροπία. Ε, και η δεξιά ήδη έσπευσε να χαιρετήσει αυτήν την πορεία. Άρα παραπάνω λιτότητα. Και τώρα, φυσικά δεν τα έχουμε αγοράσει όλα ακόμα, ναι. Και σα συγχαίρουμε ε, που μιλάτε για τον φόρ, για τα πλαστικά, για το διοξίδιο του άνθρακα, για του ε, νέου ίδιους πόρου που έχουν αξιέπαινου οικολογικού πόρου και θα απαλύνουν λίγο το βάρο των κρατών μέλων ταυτόχρονα αρνείστε ε, τους υπερεκατομμυριούχους και ε, ε, όσους επωφελήθηκαν από την κρίση όπως τα σούπερ μάρκετ για παράδειγμα που ανέβασαν το τζίρο τους κατά 35% αρνείστε αυτούς να τους φορολογήσετε και επιτρέπετε τα κράτη που πλήγονται περισσότερο να ουσιαστικά να μην έχουν μεγαλύτερη ενίσχυση. Δεν αλλάζει τίποτα στην παγκόσμια εξίσωση γιατί πάντα τα κράτη ε, που είναι πιο αδύναμα θα πληρώνουν την ύφη και άρα ο απλός ευρωπαϊκός πολίτης. Μιλάμε για 750 δις στο πλαίσιο αυτού του νέου εργαλείου, αλλά είναι παρότι κάτι καλό είναι το 1 τρίτο αυτού που είχαμε ζητήσει από την ε, δεξιά στην αριστερά πτέρυγα του Κοινοβουλίου. Και επίσης 500 ε, δις λέτε ότι είναι ε, άμεσες επιχορηγήσεις. Ε, όμως ε, κατά πάσα πιθανότητα ήδη οι πόροι που δεν είπατε ακριβώ για ποιο ποσό μιλάμε ακριβώ, μάλλον δεν θα είναι αρκετοί. Ε, οπότε θα χρειαστεί να χρεωθούν ακόμη περισσότερο τα κράτη-μέλη ώστε μέσω του ευρωπαϊκού προπολογισμού ε, να καλύψουν. Και τα λέτε ε, αυτό τα κονδύλια νέα γενιά. Μα είναι ηρωνικό αυτό. Γιατί από αυτού, από του νέου, από τη νέα γενιά ζητάτε να πληρώσει το λογαριασμό. Επομένω, πίσω από όλα αυτά κρύβεται ένα κεντρικό εργαλείο που υποτίθεται ότι θα μα οδηγήσει σε μικρότερη λιτότητα, αλλά τελικά ε, θα έχουμε άλλες ε, εξελίξεις. Το θέμα είναι να είχαμε ε, άλλα μέτρα όπως είναι τα ομόλογα στενικές για να μην έχουμε την εξάρτηση των χωρών από την τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Θέλουμε να καταπολεμήσουμε τις ανισότητες όμως. Σήμερα πώς μιλάμε για τον τρόπο με τον οποίο θα έχουμε νέα ε, δημοσιονομική ισορροπία και ταυτόχρονα ε, θέλουμε αλληλεγγύη και πρόοδο. Προς τα πού οδηγόμαστε. Δεν μπορούμε να καταργούμε θέσει εργασία όπω η Ρενό. Δεν πρέπει να παίρνετε ένα φράγκο η εταιρεία αυτή. Ούτε άλλε προ ε, τα στευτικές πρακτικές. washing είναι αυτό που γίνεται. Σώζουμε ε, τις ε, αναχρονιστικές βιομηχανίες ε, ουσιαστικά. Αντίθετα θα έπρεπε να προωθήσουμε οικολογικές εναλλακτικές, ε, την επιμερισμό του πλούτου, να παγώσει η πληρωμή να έχουν μια οικολογική πορεία. Εμείς αυτό που προτείνουμε ακριβώς είναι μια άλλη κατεύθυνση, ένας άλλος δρόμος. Θέλουμε ριζικό μετασχηματισμό του μοντέλου που έχουμε αυτή τη στιγμή για να βγούμε από την κρίση και να κάνουμε τις κοινωνίες μας πιο ανθεκτικές απέναντι στους μελλοντικού κραδασμούς. Ε, σας ευχαριστώ. Άντιν Όλφη, για τους μη εγγεγραμμένους παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτά τα οποία ακούμε μέχρι στιγμής ε, δεν μας δίνουν μεγάλες ελπίδες. Μιλάμε για ε, μεταφορές ε, σε ένα ταμείο χαμένο το οποίο θα φτιαχτεί από δάνεια. Πάρα πολλά αυτά τα οποία μας λέτε για μια πράσινη μετάβαση και ψηφιακή την οποία εμείς ζητάμε εδώ καιρό αλλά τώρα ξεκινούν τα δύσκολα. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα στο Συμβούλιο όπου κάποιες ε, χώρες ε, προωθούν πολιτικές λιτότητας. Λοιπόν, οι χώρε αυτές δεν πρέπει να λέγονται χώρε συνεπεί και οικονομε, αλλά εγωιστικέ, λοιπόν. Θα πρέπει να ξεκινήσουν ξανά οι επενδύσει. Γι' αυτό το λόγο το κίνημα των πέντε αστέρων αναμένει μια σοβαρή στήριξη από την ε, Ευρώπη. Εδώ και δεκαετίες η Ευρώπη αρνείται να αλλάξει τρόπο δράσης ε, και δυστυχώς και σε μια καταστροφή όπως αυτή την οποία ζήσαμε είδαμε ε, να εμφανίζεται το αντίθετο από αυτό το οποίο θέλαμε, δηλαδή το ευρωπαϊκό πνεύμα της ελληνικής Θα γράψουμε ιστορία, ας το δούμε. Σας ευχαριστώ κύριε Αντινόλφη. Κοιτάξτε, ε, λυπούμε. Δυστυχώ πρέπει να σεβαστούμε τους κανόνες της απόστασης. Είναι υποχρεωτικό. Οπότε Ε, να με συγχωρείτε αν ε, σας υποδεικνύουν άλλες θέσεις οι κλητήρες. Υπάρχουν δύο-τρεις αίθουσε για όλους τους βουλευτέ που θέλουν να παρακολουθήσουν. Βεβαίω οι ομιλητές ε, λογικό είναι να είναι παρόντες εδώ στην Ολομέλεια. Μουρεσάν, κύριε Μουρεσάν, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε Φοντερ Λάιν, καλώ ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ευχαριστούμε για την πρότασή σα. Αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα είναι πολύ σημαντική μέρα. Είναι σπουδαία μέρα γιατί οι πολίτε τη Ευρώπη περιμένουν βοήθεια και στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σήμερα μπορεί να του πούμε έρχεται η βοήθεια, είναι στο δρόμο, γιατί περιμένουμε την υλοποίηση του πακέτου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόκειται για ένα νέο μηχανισμό και η στήριξή του θα είναι συγκεκριμένη και θα κάνει τη διαφορά για τις επιχειρήσεις, τον κόσμο, τις περιφέρειες και τις χώρες. Ποια θα είναι τώρα τα επόμενα βήματα. Σήμερα είναι μόνο η αρχή. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε το καλύτερο δυνατό πακέτο ανάκαμψης. Και γι' αυτό θα πρέπει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εμπλακεί πλήρω αυτή την εκπόνηση τη δέσμη μέτρων. Οι συνάδελφοι εδώ προέρχονται από όλε τι περιφέρειε Ευρώπη και έχουν άμεση και μόνιμη επαφή με του πολίτε Ευρώπη. Γνωρίζουν τι ανάγκε του επιτόπου. Τι χρειάζονται τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσει, ο κόσμο. Και γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να αναμειχθεί πλήρω στον τρόπο δρομολόγηση και δαπάνη των κονδυλίων του πακέτου ανάκαμψη και τη επιστροφή κάποιων κονδυλίων γιατί η ανάμειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα εξασφαλίσει ε, το πακέτο αυτό ανάκαμψη να είναι το καλύτερο δυνατό που μπορούμε να διαμορφώσουμε από κοινού. Αυτή η δεσμή μέτρων θα επηρεάσει το μέλλον των πολιτών. Και γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που εκπροσωπεί του πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εμπλακεί πλήρω στην διαδικασία αυτή. Επίση θα πρέπει να έχουμε μια συνολική εικόνα. Η πρόεδρο Φοντερ Λάιν μίλησε για τον προπολογισμό που θα πρέπει να είναι ενιαίο. Θα πρέπει να έχουμε φυσικά το σχέδιο ανάπτυξη για να βοηθήσουμε την οικονομία και τον κόσμο να εξέλθει από την κρίση, αλλά α μην ξεχνούμε και τι παλιέ μα προτεραιότητε του κοινοτικού προπολογισμού. Α μην ξεχνούμε του γεωργού μα, του αγρότε μα, του ε, φοιτητέ μα. Α μην ξεχνούμε και τι νέε μα προτεραιότητε, την πράσινη συμφωνία, την ασφάλεια των πολιτών, την ψηφιοποίηση. Θα πρέπει να έχουμε αρκετά αποθεματικά για να ανταποκριθούμε και να αντιμετωπίσουμε απρόβλεπτε κρίσει που θα ε, σκύψουν στο μέλλον και προσβλέπουμε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αυτή τη βάση και περιμένουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεργαστεί σε αυτή τη βάση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ, Μπενιφέη, για ένα λεπτό. Ναι, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρία Φάντελαιν, σήμερα ο κόσμος κοιτάει εδώ για να δει εάν η ένωσή μα η οποία έχει βασιστεί στο κράτος δικαίου και σε ένα μοναδικό κοινωνικό μοντέλο προϊόν 10 ετιών θα μπορέσει να επιζήσει από την κρίση αυτή. Η πρότασή σας είναι φιλόδοξη. Είναι επαρκής και ανταποκρίνεται στο μέτρο της ε, κρίσης. 750 δισεκατομμύρια εκ των οποίων ένα σημαντικό κομμάτι για την ανάκαμψη επιτέλους δίνει μια σημαντική απάντηση στην έκκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για μια κοινή αλληλεγγύη την οποία ζητάμε σε αυτήν την αίθουσα. Θα επαναλάβω αυτό το οποίο είπε ο κύριος Σασόλη, ο πρόεδρος. Εμείς θα σας στηρίξουμε για να διατηρηθεί αυτή η φιλοδοξία. Λοιπόν, οι κυβερνήσει τώρα πρέπει να είναι συνεπίστα, Θα πρέπει να στηριχθεί μια νέα γενιά Ευρωπαίων. Οπότε πρέπει να κινηθούμε γρήγορα με τρόπο απλό. Οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ. ΑΙΕ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, κύριε και κύριοι, πρόκειται για μια σημαντική πρόοδο, αλλά θα, είμαι, θα τα πω ομά πράγματα και άμεσα. Πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα που θα χρηματοδοτήσουν την ανάκαμψη, τα ξέρουμε. Στην Google, στην Amazon, στο Facebook, εκεί είναι αυτά τα λεφτά. Σε όλες αυτές τις πολυεθνικές ε, που χρησιμοποιούν επιθετικό φιλικό σχεδιασμό πρέπει να επιμεριστούν το αυτό Το ίδιο για τι μεγάλε κινεζικέ επιχειρήσεις που μολύνουν και δεν τηρούν τα δικά μας πρότυπα. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το όπλο. Ε, δεν θα πρέπει το 2020, αλλά τώρα να χρησιμοποιήσουμε το όπλο των ιδιών πόρων. Και όταν θα συλλεγούν αυτά τα χρήματα για να χρησιμοποιηθούν εκεί που πρέπει. Θέλουμε να δοθεί νέα ανάσα, να έχουμε καθαρά οχήματα, ε, μονομένα ε, κτίρια, επιστροφή με τεστημένων επιχείρησεων κτλ. Ο ιό δεν διαδίδει το θάνατο μόνο, αλλά και την απελπισία, την απόγνωση. Θα πρέπει να ε, σταματήσουν να νιώθουν απεγνωσμένοι Ευρώπαιοι, αλλά φιλόδοξοι, για να, το, να αισιόδοξοι. Για να το πετύχουμε αυτό πρέπει να σα δώσουμε μια ακόμη ανάσα. Σας ευχαριστώ πάντσα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλό απόγευμα κυρία Φόντερ Λάιν. Αυτό το οποίο μας ε, παρουσιάζεται σήμερα το παρουσίασαν την προηγούμενη εβδομάδα με άλλο όνομα ο κύριος Μακρόν με την κυρία Μέρκελ, αποδεικνύοντας ακόμη μια φορά πως η Κομισιόν ακολουθεί το γαλλογερμανικό άξονα. Λοιπόν, εμείς οι Ιταλοί είδαμε αρκετή φιλοδοξία από την κυβέρνηση Κόντε, αλλά δεν έγιναν αρκετά πράγματα. Υπήρχε το ο, Ταμείο Ένταξη. αλλά οπότε θα μου επιτρέψετε μια κάποια δυσπιστία. Για να χρηματοδοτηθεί αυτό το ταμείο θα επιβληθούν νέοι φόροι. Νέοι φόροι οι οποίοι πάλι θα πέσουν στις μικρές επιχειρήσεις και τους καταναλωτές και θα ε, επιδεινώσουν την κρίση την οποία θέλετε να καταπολεμήσετε. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα επίσης ε, πρέπει να λάβουν υπόψη και τον τουρισμό, ο οποίος είναι απαραίτητος για την οικονομία πολλών ε, χωρών. Και βεβαίως ε, βλέπουμε το τι γίνεται και από τους Ολλανδούς και άλλους. Εν τω μεταξύ, βεβαίως η ευρωπαϊκή οικονομία πεθαίνει από τον κορονοϊό ή από την γραφειοκρατία. Λοιπόν, ε, μπορεί εσείς να λέτε ότι υπάρχουν λαϊκιστές, αλλά είναι απλά η καρπή των όσων εσείς σπέρνετε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρότασή τη. Γιατί δημιουργεί κάποιο χώρο για το επενδυτικό σχέδιο. Το επενδυτικό σχέδιο που χρειάζεται πάση θυσία η Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα πρέπει να προέλθει από την Ευρώπη, όχι μόνο από τα κράτη-μέλη. Γιατί αν το αφήσουμε στα κράτη-μέλη, θα έχουμε ένα, ε, μια αύξηση των ανισορροπιών στην ε, εσωτερική αγορά. Κάτι που υπάρχει ήδη. Αυτή τη στιγμή η Γερμανία δίνει τι μισέ κρατικέ ενισχύσει. Φαίνεται η ανισορροπία λοιπόν. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό επενδυτικό σχέδιο. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ευχαριστώ. Επίσης, ελπίζω και οι άλλες πολιτικές ε, οικογένειες και η κυβέρνησή μου στην Ολλανδία θα συνειδητοποιήσουν πόσο χρειαζόμαστε οπωσδήποτε ένα νέο τέτοιο επενδυτικό σχέδιο. Αλλά αυτό σημαίνει για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι οι επενδύσεις θα χρησιμοποιηθούν για την ψηφιοποίηση και την πράσινη συμφωνία. Γιατί υπάρχει στη θεωρία στα λόγια, αλλά θα πρέπει να τα εφαρμόσουμε και στα έργα και εμπράκτος. Επίσης, μιλούμε για 750 δις αλλά στις κρατικές ενισχύσεις μιλάμε για πάνω από 2-3. Και εκεί η βοήθεια δεν συνοδεύεται από όρους. Η Επίτροπος Φεστάγκερ είπε να βάλουμε όρους και στις κρατικές ενισχύσεις γιατί χρειάζονται όροι και για τις εθνικές επενδύσεις και για τις κρατικές ενισχύσεις, γιατί εκεί θα αποκαταστήσουμε την ισορροπία στην οικονομία. Η κυρία Σίντουο, για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται σήμερα την ελληνική και οι Ευρωπαίοι πολίτε χρειάζονται ελπίδα. Με ικανοποίηση άκουσα την παρουσίαση τη Πρόεδρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μίλησε για περισσότερα κονδύλια, για ένα δαψιλό ταμείο. Αλλά θα πρέπει να εξετάσουμε και τις λεπτομέρειες, γιατί πολλοί μίλησαν για την αύξηση των ιδίων πόρων και νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή να ξεκινήσουμε την καταπολέμηση των φορολογικών απατών και της φορο... φοροδιαφυγής. Επίσης, η Πρόεδρος είπε ότι ήρθε η στιγμή που θα πρέπει να απομακρυνθούμε από τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα. Και πιστεύω ότι τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καθοδηγηθεί κυρίω από τι αρχέ τη ε, συνθήκη, των συνθήκων και θα δείξει αλληλεγγύη. Θα λάβει υπόψη την κατάσταση σε όλε τι χώρε μέλη και θα αντιμετωπίσει ε, ισότιμα τα κράτη-μέλη ε, λαμβάνοντα υπόψη τι ανάγκε του. Γιατί οι πολίτε ε, χρειάζονται δουλειά και ελπίδα και είμαστε υποχρεωμένοι, έχουμε το καθήκον να του το δώσουμε. Πρέγκο, Μάρτον, um, <clears throat> Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πέραν τη ουσία, είναι πραγματικά τρομερό που σε μια κρίσιμη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπονεί μια συμφωνία και κλεισμένο των θυρών επικρίνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση για αδιαφάνεια και έχουν δίκιο. Γιατί αν θέλει να φαίνεται δημοκρατική η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να το κάνει και στην πράξη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και στην τελευταία συμφωνία του Ιουνίου του 2018, Μακρόν και Μέρκελ για την ε, Δημοσιονομική ε, Ένωση, Φορολογική Ένωση, ελπίζω η σημερινή ε, συμφωνία να είναι καλύτερη, γιατί η συμφωνία του 2018 εξαφανίστηκε. Και δεν ακούσαμε τίποτα μετά τις διακηρύξεις. Ελπίζουμε πάντως αυτό το πακέτο, αυτή η δεσμή μέτρων θα εφαρμοστεί αποτελεσματικά, αλλά έχω κάποιες ε, ανησυχίες. Φοβάμαι ότι αυτό το Ταμείο των 500 δισεκατομμυρίων να μην λειτουργήσει ως ευρωομόλογο, δηλαδή να μην μεταφέρει ε, χρέη από το εθνικό επίπεδο στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί έτσι απλώς θα προσθέσει ε, στο αβάσταχτο ε, φορτίο του χρέους πολλών ε, χωρών που ήδη έχει καταποντήσει τις οικονομίες τους. Θέλω και εγγυήσει σε αυτό το σχέδιο ανάκαμψης, ώστε τα κονδύλια να μην πάνε στους μεγάλους ομίλους και τις πολυεθνικές, αλλά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί αυτές είναι η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας. Κύριε Αντελάνγκε, για δύο λεπτά παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, Επίτροπη. Να μιλήσω Ολλανδικά γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό. Θα ήθελα να καλωσορίσω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, πρέπει να αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην τρέχουσα κρίση. Και βεβαίως ακούσαμε για τη διαφορά μεταξύ επιδοτήσεων και δανείων ε, κτλ. Αλλά καλωσορίζω αυτή την πρόταση. Και βεβαίως ε, υπάρχει και η ατμόσφαιρα η οποία δημιουργείται, γιατί όλοι στην ίδια βάρκα είμαστε. Θα πρέπει λοιπόν να βγούμε μαζί από αυτήν την κρίση. Επίσης, ακούστηκαν διάφορα για ψηφιακό φόρο, τα χαιρετίζω, αλλά για μένα το βασικό είναι ότι επιτέλους θα διατεθούν τα κονδύλια. Και αυτό το οποίο ανησυχεί είναι ότι τώρα μπαίνουμε σε χρέος, είναι αναπόφευκτο σε αυτήν την κρίση, αλλά είναι σαφές, ασαφές το πώς θα πληρωθεί και η ανησυχία μου είναι ότι αν δεν έχουμε ίδιους πόρου. γιατί εάν είναι ένα κράτο μέλο κατά δεν θα έχουμε, τελικά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον ευρωπαϊκό προπολογισμό για να ξεπληρώσουμε αυτό το χρέο με λιγότερα λεφτά για να ασκήσουμε πολιτική. Οπότε εγώ θα ήθελα να δω μια πραγματική δέσμευση από το Συμβούλιο ότι θα έχουμε ίδιους πόρους ή ότι θα ξεκινήσει ένα σχέδιο αποπληρωνής ήδη από το τρέχον ΠΔΠ. Πρέπει να είναι σαφές αυτό για να λειτουργήσει αυτό το πρόγραμμα. Και να πω κάτι στην κυρία Γκαρσία Πέρε. Μόλι είπα στα Ολλανδικά, στη γλώσσα μου, γιατί είναι σημαντικό, ότι πρέπει όλοι μαζί να στηρίξουμε αυτή την πρόταση ότι όλοι στην ίδια βάρκα είμαστε. Αλλά εάν προτείνεται να γίνει αυτό το θέμα 23 εναντίον 4 δεν θα επιτύχουμε. Θα εξωθήσετε αυτές τις τέσσερις χώρες στα χέρια της άκρας δεξιάς. Εάν πείτε να το κάνουμε χωρίς ομοφωνία. Να βασίζεστε στις φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις αυτών των χωρών και σε εμένα, αλλά πρέπει να το κάνουμε από κοινού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Γκάιερ. Γιάννης, για ένα λεπτό. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύρια Πρόεδρε Φόντερ Λάιν. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το ότι ήρθατε εδώ όταν υποβάλει το εκτελεστικό ένα σχέδιο, νομίζω καλό είναι να έρχεται να το υποβάλει στον τόπο της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας, στο Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ λοιπόν και χαιρετίζω την Κομισιόν για την πρόταση την οποία έκανε. Νομίζω έχει επαρκή ε, έκταση και στόχους. Βεβαίως με απογοητεύεται λίγο γιατί δεν προτείνα τίποτα για τους ίδιους πόρους. Γίνονται διάφορες καλές προτάσεις, οποίες όλοι έχουμε συζητήσει, αλλά όλα είναι σε υποθετικό λόγο. Ε, λοιπόν, βλέποντας την κατάσταση στο Συμβούλιο, νομίζω ότι έχει σχέση με τις, ε, τους σχετισμούς εκεί μέσα. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω ποιους ίδιους πόρους θέλετε εσείς να δείτε και τι προτείνετε σε Συμβούλιο και Κοινοβούλιο. Θα έχετε οπωσδήποτε την στήριξή μας. Καλό λοιπόν θα ήταν να μας πείτε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι φρενάρουν. Ένα άλλο το οποίο με ανισχύει είναι από πού θα βρούμε τα λεφτά. Πρέπει να είναι και ξεκάθαρε οι προτεραιοτητε καινοτομια καινοτομία, κοινωνικό-οικολογικός μετασχηματισμός, αυτά. Λοιπόν, δεν ε, βλέπω αρκετά πράγματα για αυτές τις προτεραιότητε. Σας ευχαριστώ. Κάνο για ένα λεπτό. Τις μέρες αυτές οι Ευρωπαίοι πολίτε βγαίνουν με προσοχή από τα σπίτια του. δείξαμε υπευθυνότητα και βελτιώθηκε η υγειονομική κατάσταση. Όμω ε, η οικονομική κατάσταση είναι σαν την κόλαση του δάντη. Όσοι έχουν ένα μικρό μαγαζί ή δουλεύουν κάπου, δεν ξέρουν αν στο τέλο του μήνα θα έχουν ακόμη τη θέση εργασία του. Και πολλοί εκατομμύρια Ευρωπαίοι φοβούνται για το μέλλον του. Χαιρόμαστε που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άκουσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα αιτήματά του που διατυπώθηκαν πριν από δύο εβδομάδε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκδώσει χρέο ε, από κοινού για να στηρίξει ένα σχέδιο οικονομική ανάκαμψη. Επίση, θα πρέπει να απευθύνω μια έκκληση ευθύνη και υπευθυνότητα και προ τα κράτη-μέλη. Το σχέδιο αυτό επήγει. Κάθε μέρα που περνάει πάνω από 2.000 επιχειρήσει κατεβάζουν λουκέτο, χρεοκοπούν στη χώρα μου. Κάθε μέρα που χάνουμε σε στήρες συζητήσει ε, θα χάνουμε θέσει απασχόλησης και θα καταστρέφουμε ζωές. Θα πρέπει τώρα να δράσουμε και επίσης να κάνουμε πραγματικότητα, να δώσουμε σάρκα και οστά σε αυτό το σχέδιο, γιατί αυτό περιμένουν οι Ευρωπαίοι και δεν θα πρέπει να τους απογοητεύσουμε. Αυτή είναι η στιγμή της ε, αλήθειας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το μέλλον της εξαρτησίας. Σας ευχαριστώ, Ζουβάν, για ένα λεπτό. Σα ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Μας αναφέρατε ε, πάρα πολλά ε, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, τα οποία ουσιαστικά είναι η αλυσίδα ε, με την, με την οποία θα δέσετε το πόδι της νέας γενιάς. Μιλάμε ε, ουσιαστικά ε, για ένα, μια ευρωπαϊκή ε, οικονομία και πολλά άλλα προγράμματα. Αυτό το σχέδιο όμως νομίζω ότι θέλει να πετύχει κάτι που δεν γίνεται, δηλαδή την επιστροφή στο παρελθόν. Αυτό δεν γίνεται και πρέπει να ετοιμάσουμε τον κόσμο για το μέλλον, σε έναν κόσμο που θα ζουν ασφαλείς οι πολίτες. Αυτό λοιπόν τον κόσμο που θέλουμε να ετοιμάσουμε για το μέλλον, εκεί η ποιότητα θα μετρά περισσότερο από την ποσότητα. Η εσωτερική αγορά, η προτίμηση των προϊόντων προέλευσης θα πρέπει να είναι εγγυημένη. Θέλουμε έναν κόσμο αλληλεγγύης Πρέπει να πάψουμε να σκεφτόμαστε με όρους ε, άκρατης και άναρχης ανάπτυξης. Θα πρέπει να, να προσέξουμε ε, μήπως στο τέλος ε, έχουμε τους επόμενους μήνες κατάρρευση οικονομική και κοινωνική. Ευχαριστώ πολύ. Καρέμνα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη είναι αναγκαία απέναντι σε αυτή την άνευ προηγουμένου κρίση, αμοιβαιοποίηση λοιπόν ενισχύσεων και σεβασμό στο Ευρωκοινοβούλιο. Όλα αυτά είναι θετικά. Θα έλεγα ότι είναι και ιστορικά. Αρκεί να οι προτάσει αυτέ από περισσότερη φιλοδοξία και αν είχαμε εγγυήσει ότι θα προχωρήσουμε σε μετασχηματισμό τη οικονομία, σε οικολογικό μετασχηματισμό ε, και να μην έχουμε μια φυγή προ τα εμπρό ε, απλά. Ε, θεωρώ ότι θα μπορούσε να είναι πιο φιλόδοξο φιλόδοξο το πρόγραμμά σας, ε, διότι δεν ε, θα βοηθηθούν όλοι οι συμπολίτες, ούτε αρκούν αυτά τα μέτρα για να αντιμετωπίσουμε την εξαφάνιση των ειδών, να προστατεύσουμε το κλίμα μέσω της ε, Συμφωνίας του Παρίσι κτλ. Εγώ, σαν καλό Γάλλος, δεν εμπιστεύομαι τα λόγια, θέλω έργα. Είπατε ότι με την αδράνεια θα μας κοστίσει πολύ περισσότερο. Γιατί λοιπόν να μην αναλάβουμε ήδη από τώρα μαζικά δράση, διότι πεθαίνουμε από τον αέρα που αναπνέουμε από το νερό που πίνουμε. Παραμορφώνεται το πρόσωπο της Ευρώπης με τις μάσκες που φορούμε σήμερα. Τι μέλλον θέλουμε, αν ακούσουμε οικολόγους, ε, νοσηλευτές, ε, νεολαία, δεν είναι καλύτερα από το να, μιλά, να μιλάνε μόνο αυτοί ε, που μιλούν για κρίση και για λιτότητα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Έπινγκ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ένα πολιτικό πραξικόπημα. Το θέμα δεν είναι ο κορονοϊός, αλλά η εξουσία στην Ευρωζώνη και στις Βρυξέλλες. Ε, βρισκόμαστε στο κατόφλι μιας ένωσης μεταφορών, η οποία δεν θα μπορεί να αναστραφεί πλέον, κυρία Φόντερ Λάιν. Ακόμα τα σχέδιά σας δεν έχουν περάσει βέτο υπάρχουν από 27 κράτη-μέλη για τα δισεκατομμύρια τα οποία προτείνεται, για τον νέο προϋπολογισμό και τους ε, φόρους και για αυτά τα οποία προτείνεται, τα οποία αυτή τη στιγμή αντιβαίνει το άρθρο 311 της Συνθήκη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας ίκαρος ο οποίος κατευθύνεται απευθείας στον ήλιο. Υπάρχει λοιπόν μια διαδικασία η οποία θα πρέπει να περάσει από 50 κοινοβούλια. Θα πρέπει να γίνει η συζήτηση αυτή με τους ανθρώπους οι οποίοι θα πρέπει να πληρώσουν. Και ήδη ένας Γερμανός καθηγητής έχει προσφύγει στο Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο. Θα το έκανα εγώ, δυστυχώς δεν είμαι Γερμανός καθηγητής. Σας ευχαριστώ. Ε, κύριε Πούτζεμον, για ένα λεπτό. Ε, η Ευρώπη ε, καθορίζεται ως πολιτικό σχέδιο από την απάντηση και την αντιμετώπιση των κρίσεων. Πολλοί πολίτες έχουν πολύ κακές αναμνήσεις από το πώς χειριστήκαμε την τελευταία χρηματοπιστωτική χρήση, την κρίση. Γιατί ε, ενοχοποιήθηκαν από τα έκτροπα των κυβερνήσεων και την ανικανότητα να προγραμματίσει ε, κάποιες σημαντικές αλλαγές. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε επανάληψη αυτού του λάθους. Θα πρέπει να δράξουμε αυτή την ευκαιρία που έχει η Ευρώπη με την Ευρωπαϊκή Ένωση της επόμενης γενιάς ε, για να συνεργαστούμε απευθείας με τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, να ξεπεράσουμε εθνικά σύνορα, να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο μητροπολιτικών περιοχών και περιφερειών για να μπορούσαμε ε, να αντιδράσουμε άμεσα και να είμαστε κοντά στους πολίτες. Θα πρέπει να επιλέξουμε. Και η Ευρώπη ως ε, μεγάλος διαχειριστής ε, κάποιων παλιών χωρών που είναι ανίκανες να αντιμετωπίσουν το μέλλον, τέτοια θα είναι η Ευρώπη ή θα είναι η Ευρώπη ε, που θα συνεργάζεται με τους πολίτες, που θα έχει ισοτιμία δικαιωμάτων και ελευθεριών και θα κινηθεί προς μια κοινωνική και δημοκρατική πρόοδο η Next Generation Europe, αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση επόμενη γενιά, είναι το επόμενο μήνα. Συνεχίστε χωρί καμία χρονοτριβή. Ο κύριο Κονσάλε Πόν, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Βρισκόμαστε σε μια αποφασιστική στιγμή, σε μια καμπή. Ή θα είμαστε φιλόδοξοι ή δεν θα επιβιώσουμε. Αυτό το σχέδιο των 750 δισεκατομμυρίων ευρώ που μα παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι φιλόδοξο και γι' αυτό δημιουργεί ελπίδε αλλά έχουμε πολύ δρόμο ακόμη μπροστά μα. Καταρχήν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετέχει στη χάραξη του σχεδίου ανάκαμψη. Ε, πέραν αυτού του οικονομικού σχεδίου Μάρσαλ, η Ευρώπη χρειάζεται και ένα δημοκρατικό σχέδιο Μάρσαλ. Δηλαδή, το κράτο δικαίου και οι αξίε μα ε, θα πρέπει να τύχουν υποστήριξη με την ίδια πυγμή που υποστηρίζουμε και το κοινό μα νόμισμα. Επίση, θα πρέπει να έχουμε ισότιμη και ακριβωδίκη κατανομή των κονδυλίων, να φτάνουν στου πολίτε, γιατί τα δισεκατομμύρια που αναγγέλουμε σήμερα θα είναι πραγματικά, αλλά το θέμα είναι ότι ε, όταν λέμε τρισεκατομμύρια, οι πολίτες ε, δεν μας πιστεύουν, γιατί πολλές φορές αυτά τα νούμερα δεν σημαίνουν τίποτα για αυτούς. Επίσης, θα πρέπει να διατεθούν τα κονδύλια το συντομότερο δυνατό. Εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούν να περιμένουν γιατί η χρεοκοπία θα σκοτώσει πολύ περισσότερους από τον ιό, από τον κορονοϊό. Επίσης, δεν έχουμε διαφορετικέ ανάγκε, αλλά τώρα έχουμε περισσότερε ανάγκε να ληφθεί υπόψη στον προπολογισμό. Επίση, το ταμείο αυτό δεν θα πρέπει να είναι άλοθη για τι πολιτικέ των κακών κυβερνήσεων. Γιατί αν ποτίσουμε τον λαϊκισμό, ε, το φυτό αυτό θα γιγαντωθεί. Επίσης, 27 είναι οι χώρες που βάζουν χρήματα και που λαμβάνουν χρήματα. Α μην γελιόμαστε. Τα χρήματα δεν είναι ουρανοκατέβατα. Αργά ή γρήγορα θα τα βάλουν οι πολίτες από την τσέπη του. Οπότε θα πρέπει να σκεφτούμε τους πολίτες, όχι τις κυβερνήσεις. Είναι η στιγμή να δείξει την πυγμή του το κοινωνικό κράτος. Επίση το δημοσιονομικό πλαίσιο δεν θα πρέπει να διακυβεύσει το επόμενο πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο. Γιατί στη τελική ανάλυση ε, οι εθνικές κυβερνήσεις θα εγκρίνουν το ΠΔΠ. Τέλος, η οικονομία δεν είναι μόνο νούμερα. Η οικονομία είναι και εμπιστοσύνη. Μιλούμε για ανθρώπους, για ανθρώπινα πλάσματα. Μιλούμε για τη ζωή όλων των συμπολιτών μας. Όχι για τους πολιτικούς που μας διακυβερνούν. Ευχαριστώ. Έστεμπαν. Φερνάντες, Γιώνας, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ιστορική σημερινή ημέρα. Διότι σίγουρα μπορεί να αποτελέσει την αλλαγή, ε, μια αμετάκλητη ριζική αλλαγή στην ε, ευρωπαϊκή οικοδόμηση που θα προσωμιάζει με την θέση σε ισχύ του κοινού νομίσματος. Αυτή η έκδοση κοινού χρέου ε, συνεπάγεται μια ιστορική αλλαγή στον οικονομικό και κοινωνικό σχεδιασμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα βήμα για το οποίο εδώ και δεκαετίε εργαζόμαστε και σήμερα έχουμε μια πρόταση από αυτήν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προ αυτή ακριβώ την κατεύθυνση. Πιστεύω πω η πρόταση ε, αυτή τη ανακοίνωση για αυτόν τον ε, για αυτό το νέο ταμείο ε, είναι μια στεναρή, στιβαρή, στέρεα πρόταση που πρέπει να μελετηθεί βέβαια σοβαρά γιατί ακόμα δεν είχαμε τη δυνατότητα να μελετήσουμε όλε τι λεπτομέρειε όμω δράτω με τις ευκαιρίε για να συγχαρώ το Συμβούλιο ε, και για να ζητή, την Κομισιόν και για να ζητήσω από το Συμβούλιο και από τα κράτη-μέλη να συνδράμουν ώστε να γίνει αυτό το ιστορικό βήμα προ όφελο όλων των Ευρωπαίων. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ναι, ευχαριστώ. Τάσμανι για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ναι, εντωμέσω αυτής της ε, υγειονομικής κρίσης ανέφερε προηγουμένου κανείς δεν έχει μείνει ανεπηρέαστος. Ο κόσμος αρρωσταίνει, χάνει τους οικείους του, βλέπει τις επιχειρήσεις να υποφέρουν, χάνει τη δουλειά του. Ο κόσμος λοιπόν θα πρέπει να αναλογιστεί τα πράγματα, να σκεφτεί τι είναι σημαντικό, ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητές μας. Όπως και εμείς πρέπει να αξιολογήσουμε ξανά τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Ε, αντιμετωπίζουμε αυτές τις προκλήσεις και ξέρουμε ότι έχουμε και άλλες προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε. Ο κόσμος αναμένει από εμά μία ενιαία απάντηση. Να είμαστε υπόλογοι και να μην με δώσουμε το βάρος στις επόμενες γενιές. Για να το επιτύχουμε αυτό πρέπει να έχουμε ως προτεραιότητα τα σημαντικά, να δούμε πώς μπορούμε να εστιάσουμε τις οικονομίες μας και να τις μεταρρυθμίσουμε για να βγουν ισχυρότερες αλλά από κοινού. Όπως και οι πολίτες μας προσπαθούν να προσαρμοστούν σε αυτήν την κρίση. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και εμείς για να μπορούμε να ανακάμψουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Χάιντερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύρια Πρόεδρε. Στην Ευρώπη εκατομμύρια άνθρωποι χάνουν τις δουλειές τους, δεν ξέρουν πώς θα θρέψουν τις οικογένειές τους, ενώ εκατομμύρια άνθρωποι φοβούνται για το ψωμί τους. Έρχεται εδώ πέρα το Κοινοβούλιο να συνεδριάσει κοστίζοντας χιλιάδες ευρώ. Γιατί? Όχι για τον προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός δεν υπάρχει. Είναι ένας ε, προϋπολογισμός φαντασμά. Όχι, δεν συζητάμε γι' αυτό έχουμε μία πρόεδρο της Κομισιόν η οποία ήρθε εδώ για να μας κάνει προπαγάνδα. Αυτή ήταν η σημερινή παράσταση της κυρίας ε, Φοντελαϊν. Και μιλάμε για χιλιάδες εκατομμύρια ευρώ τα οποία πετάγονται εν το μέσο της μεγαλύτερης κρίσης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έχουμε αναδιανομή από βορρά προς νότο και δεύτερον έχουμε το όνομα όλων των ευρωκρατών να έχουν φόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μην ζητάνε την άδεια των Εθνικών Κοινοβουλίων. Αυτό είναι ο στόχο. Δεν θέλει να καταπολεμήσει την κρίση. Θέλει να εκμεταλλευτεί την κρίση για να επιτύχει τον στόχο ενό υπερκράτου των Βρυξελών. Σα ευχαριστώ. Ουρτασούν. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Το πακέτο είναι πολύ σημαντικό και πολύ σημαντικό άλμα υπέρ της ολοκλήρωσης της Ευρωζώνης. Και είναι σημαντικό πολιτικό μήνυμα προ του Ευρωπαίου πολίτε. Από κοινού θα χρεωθούμε για να αντιμετωπίσουμε από κοινού την κρίση. Φυσικά θα θέλαμε κάτι περισσότερο, μια δέσμη μέτρων με μεγαλύτερο μακροοικονομικό αντίκτυπο. Αλλά είναι το ελάχιστο για να διασώσουμε την ε, εσωτερική αγορά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το μέλλον των εκατομμύριων Ευρωπαίων πολιτών δεν μπορεί να γίνει όμοιρος στις ε, επιθυμίες τεσσάρων κυβερνήσεων που δεν ε, βρίσκονται στο ύψος των περιστάσεων. Επίσης, θα ήθελα να πω τρία ε, σχόλια. Καταρχήν, και η ψηφιακό μετασχηματισμό και ο οικολογικό μετασχηματισμό είναι σημαντικά, αλλά μην ξεχνούμε και τι κοινωνίε που έχουν πληγεί από την προηγούμενη κρίση. Επίση, θα πρέπει να εκδημοκρατήσουμε το σύστημα χάραξη των μεταρρυθμίσεων. Δεν μπορεί οι τεχνοκρατικές συστάσεις να μην υπόκεινται σε έλεγχο από τα κράτη. Επίσης, να καταπολεμήσουμε αντικοινωνικές μεταρρυθμίσεις με λιτότητα που τόσο έπληξαν τις κοινωνίες. Να έχουμε το σχέδιο ανάκαμψης και να το κάνουμε ένα χρήσιμο εργαλείο. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Φιντάντσα, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μετά από εβδομάδες ή και μήνες επιτέλους έχουμε μια ξεκάθαρη πρόταση. Αλλά Έχουμε πάρα πολλά σημεία ε, κρίσιμα. Πρώτα απ' όλα να δούμε τις συνεισφορές, γιατί 500 δισεκατομμύρια είναι ένα μήνυμα αλλά δεν φτάνουν. Δεύτερον, τα λεφτά αυτά θα πρέπει να εκταμιευθούν αμέσως ε, τους ε, επόμενους έξι μήνες, αλλιώς δεν θα κάνουμε τρίτο. Τρίτον, ο προορισμός, γιατί έχουμε πάντα τις ίδιες ιδεολογικές προτεραιότητες σαν να μην έχει υπάρξει ποτέ ο ιός. Τέταρτον, η αιρεσιμότητα. Γιατί βλέπουμε πάλι αυτά τα οποία ζητάνε οι Βρυξέλλες να κάνουμε μεταρρυθμίσεις. Και βεβαίως πέμπτο, ήδη οι πόροι, νέοι ευρωπαϊκοί φόροι δηλαδή. Θα πρέπει να σκεφτούμε πώς ένα σεντ παραπάνω φόρων επηρεάζει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Αυτά. Ευχαριστώ. Ρέγνερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Κομισιόν με την πρόταση αυτή μας δείχνει πως υπάρχει μία λύση μόνο. Περισσότερο θάρρος, περισσότερη αλληλεγγύη και περισσότερη Ευρώπη. Καμία χώρα δεν είναι απομονωμένη. Και αυτό θα ήθελα να το απευθύνω προς τους ε, τέσσερις αγωνιστικές χώρες και προς την Αυστρία. Θα πρέπει να σταματήσετε επιτέλους να σκέφτεστε μόνο την χώρα. Η Ευρώπη θα επιτύχει από κοινού ή θα αποτύχει. Θυμηθείτε τις υποσχέσεις σας κατά τη διάρκεια της ε, Προεδρίας της Αυστριακής. Μια Ευρώπη η οποία προστατεύει, η οποία προστατεύει τους άρρωστους, προστατεύει τους νέους, προστατεύει τις γυναίκες που επηρεάζονται ιδιαίτερα από αυτή την κρίση. Γι' αυτό ακριβώς ε, θα πρέπει να τηρήσουμε τις υποσχέσεις αυτές, να θα προστατεύσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Πρέπει να το κάνουμε και αυτό σημαίνει ότι τα μισά από αυτά τα κονδύλια θα πρέπει να πάνε στις γυναίκες. Οι γυναίκες, ο μισός πληθυσμός δηλαδή, να ωφεληθεί γιατί έχει πληγεί ιδιαίτερα από αυτή την κρίση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Άνε Μανσία, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ερχόμενος εδώ στο Ζάβεντον ε, είδα πως ε, κατάφερε ένας ε, οικολόγος υπουργό εδώ πέρα να κλείσει μια λωρίδα της ε, Rue de la Ήταν πάντα το όνειρό τους και τώρα βλέπουμε ότι οι διάφοροι πολιτικοί εκμεταλλεύονται την κατάσταση για τα διάφορα όνειρά τους, για το φεντεραλιστικό όνειρο εδώ πέρα. αυτά τα οποία ακούμε δηλαδή για κοινά χρέη, για προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία αποφασίζονται και κλεισμένων των θυρών ε, από τη μια μέρα στην άλλη. Η κυρία Φοντερ Λάιν μας είπε πως ε, ο κορονοϊός είναι η στιγμή της Ευρώπης. Ναι, ίσως για εσάς και για την ελίτ εδώ πέρα, αλλά για τους ε, λαούς της Ευρώπης είναι μια σκοτεινή στιγμή και πρόκειται για φοβερή επίθεση κατά των λαών, κάτι το οποίο με θλίβει. Σας ευχαριστώ για την Κομισιόν κύριος έχει τώρα τον λόγο Thank Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμοι ευρωβουλευτές, αγαπητοί συνάδελφοι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί νομίζω ότι το μήνυμα από τις περισσότερες παρεμβάσεις ε, είναι μια υποστήριξη, ένθερη υποστήριξη της προτάσεις που κατέθεσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλω να σας ευχαριστώ για την έμπνευση που μας ε, έχετε πολλές φορές προσφέρει με τα ψηφίσματά σας, με τις συζητήσεις σας ε, στις οποίες έχουμε μέχρι τώρα παραστεί για να δούμε ε, πώς μπορούμε καλύτερα να τα αποκριθούμε στα αιτήματά σας και να δείξουμε μεγαλύτερη αλληλεγγύη για να χρησιμοποιήσουμε αυτή την κρίση ως μια ευκαιρία για τον εξυγχρονισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας και για να παγιώσουμε, να εδραιώσουμε τη θέση της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο παγκόσμιο προσκήνιο ως παγκόσμιο πρωταγωνιστή. Κάναμε μια πρόταση που είναι πραγματικά πρωτάκουστη και άνευ προηγουμένη. Διότι αυτό το οποίο θέλαμε είναι το αρχικό, ε, τις αρχικές με μουσομικές πολιτικέ, να τι προσαρμόσουμε στι ε, σημερινέ ανάγκε, αλλά και γιατί αντιλαμβανόμαστε πόσο οξία είναι, ε, πόσο βαθιά είναι αυτή η οικονομική και υγειονομική κρίση. Άρα χρειαζόταν ένα νέο εργαλείο, το οποίο έχει πάρει το όνομα Next Generation EU. Ουσιαστικά μιλάμε για 1,13 ε, της πρότασης για το ΠΔΕΛΤΑΠΗ και 750 δις ε, ευρώ για το New Generation που όπως ε, ε, είχατε ζητήσει και με το ψήφισμά σα, ε, θα διατεθεί υπό μορφή επιχορηγήσεων και δανείων. Θέλω να ευχαριστήσω την ε, κυρία Πέρες, του κυρίους Μάνφρεντ Βέμπερ και Τσιόλος που υποστήριξαν αυτή την προσέγγιση κομισιών. Η επιτυχία των προτάσεων αυτών βέβαια είναι κάτι το οποίο θα κρυφθεί εκ του αποτελέσματος αν επενδυθούν τα κονδύλια αυτά στου σωστού τομεί. Και αυτό το οποίο εμείς θέλουμε ακριβώς αυτό είναι. Αντιλαμβανόμαστε απόλυτα ε, το ότι αν θέλουμε να εξυγχρονίσουμε την ευρωπαϊκή οικονομία θα πρέπει να προωθήσουμε πράσινες βιώσιμες τεχνολογίες ε, με μεγαλύτερη ψηφιοποίηση στην Ευρώπη. Και σίγουρα πρέπει να ε, διδαχθούμε από το παρελθόν για να είναι πιο ανθεκτική η ευρωπαϊκή οικονομία. Μάθαμε πόσο δύσκολο είναι να εξαρτάται κανείς από παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, από έναν και μόνο προμηθευτή για πάρα πολύ σημαντικά αγαθά, όπως το είδαμε τους τελευταίους μήνες. Αυτό λοιπόν το οποίο καταθέτουμε είναι μια πρόταση. Όχι απλά για να ξεπεράσουμε την κρίση, αλλά και για να εξυγχρονίσουμε ε, την ε, οικονομία, να δώσουμε μια κοινωνική διάσταση ε, στις πολιτικές μας και να προετοιμάσουμε τις ευρωπαϊκές κοινωνίες για την μετά την COVID-19 εποχή. Ακούσαμε παρεμβάσεις με ιδιαίτερο πάθος σε σχέση με το χρέος, σε σχέση με τους ίδιους πόρους ο κύριος Μόιτεν, κύριε Ομπρί, ο κύριο Φανόβερτβελ. Θέλω να σα πω το εξή. Εμεί έχουμε κάνει πολύ καλά ε, τη δουλειά μα. Μελετήσαμε πολύ προσεκτικά την κατάσταση και μελετήσαμε διάφορε προτάσει για του ιδίου πόρου που θα τις συζητήσουμε μαζί σα βέβαια και με τα κράτη-μέλη. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι το νέο ETS και τα έσοδα που θα έχουμε από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορία, από το θαλάσσιο, τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και των ευρωπαϊκών μεταφορών, το χρησιμοποιήσουμε αυτά τα έσοδα για να χρηματοδοτήσουμε ε, το πολιετέ ε, στο μέλλον. Επίση, θέλουμε το φόρο τη ενέα αγορά, όπω τον λέμε, ιδίω για τι εταιρείε αυτέ που αποφελούνται από το γεγονό ότι ε, λειτουργεί εύρωστα και σε τόσο μεγάλες διαστάσει τόσο μεγάλη κλίμακα είναι η αγορά. Σίγουρα θέλουμε να είναι σεβαστοί οι στόχοι της Συμφωνίας ε, του ε, Παρισίων για να έχουμε ένα μικρότερο οικολογικό αποτύπωμα και αν χρειαστεί θα έχουμε αυτό το φόρο προσαρμογής ε, που θα μπορούσε να αποτελέσει και αυτό ένα νέο πόρο, νέα έσοδα για τον ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό Και βέβαια υπάρχει το ενδεχόμενο του ψηφιακού φόρου που προσφέρει πολλές δυνατότητες. Φυσικά και θέλουμε βέβαια να υπάρξει μια γενική συμφωνία παγκόσμια στο πλαίσιο της ομάδας των 20 ή του ΟΣΑ. Αλλά αν δεν λειτουργήσει κάτι τέτοιο είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε και μόνοι μας σε αυτό το δρόμο. Για την κυρία Σίτλο και τον κύριο Ασμάνη, οι οποίοι μίλησαν για το πόσο σημαντικό είναι να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των αθέμπτων εμπορικών πρακτικών, φορολογικών πρακτικών και ε, τη φορολογική. Σίγουρα όλα αυτά θέλουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Θέλουμε σωστή εξέ, εκτέλεση του προπολογισμού και πολύ σημαντική προτεραιότητά μα βέβαια είναι και η αποφυγή τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή. Δεν κατάλαβα ακριβώ ε, όταν κάποιος μας κατηγόρησε για έλλειψη διαφάνειας, πού το ε, βρίσκεται αυτό όταν στις 12 ε, φτάνουμε να καταλήξουμε αυτές τις αποφάσεις και στη μία είμαστε εδώ για να σας τις παρουσιάσουμε. Δηλαδή είστε το πρώτο θεσμικό όργανο στο οποίο καταθέτουμε δημοσία αυτές τις προτάσεις. Ε, η πρόεδρος μας σας ανέφερε με μεγάλη λεπτομέρεια τι θέλουμε να πετύχουμε και πώς προτιθέμεθα να το πετύχουμε. Είναι μια παράδοση την οποία τηρούμε, ακολουθούμε και σεβόμαστε τον το δημοκρατικό κοινοβουλευτικό έλεγχο. Όπω και τώρα, έτσι και στο μέλλον θα συνεχίσουμε να συστούμε μαζί σα όλε αυτέ τι νομοθετικέ προτάσει που είναι πολύπλοκε και για τι οποίε χρειαζόμαστε σίγουρα τη στενή συνεργασία με εσά. Και σίγουρα θα είμαστε σε στενό συντονισμό. Υπάρχουν πολλά θέματα που έχουν να κάνουν τι κρατικέ ενισχύσει. Άκουσα αρκετέ τέτοιε ερωτήσει. Το ληστικό αντιπρόεδρο, η κυρία Φέσταγκερ, είναι γνωστό πόσο αυστηρά ε, και αντικειμενικά κρίνει όλε τι περιπτώσει και πρέπει να συμφωνήσω και εγώ μαζί σου ότι ήταν ε, πραγματικά εξαιρετική τελευταία μήνες γιατί πρώτα έπρεπε να αγωνιστούμε για να σώσουμε ζωές, για να σώσουμε ε, τις οικογένειες, τα νοικοκυριά ε, και σε ό,τι αφορά ε, την οικονομική του επιβίωση, δηλαδή να κάνουμε ό,τι έπρεπε. Αυτό ήταν η πρώτη μας προτεραιότητα. Αν, θε, αν μπορούσα να ολοκληρώσω με κάτι, αυτό θα ήταν μια έκκληση. Επειδή πραγματικά θεωρώ ότι είναι μια στιγμή μοναδική για την ιστορία της Ευρώπης, είναι ένα ορόσημο, θα πρέπει όλοι να επιδείξουμε πολιτική ηγεσία. Γι' αυτό λοιπόν θα ε, εκτιμούσουμε ιδιαίτερα την ισχυρή υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο κ. Γκονσάλεφ Πόν νομίζω το τόνισε. Χρειαζόμαστε όμω όχι την υποστήριξή σα μόνο, αλλά και τη βοήθειά σα. Να πείσετε του συμπατριώτε σα ε, στι χώρε σα. Και απευθύνομαι ε, ω προ αυτό και στο Συμβούλιο και στα κρατημέλη, διότι χρειαζόμαστε μια καλή απόφαση, μια γρήγορη απόφαση. Και βέβαια πρέπει να συνεργαστούμε στενά με όλα τα εθνικά κοινοβούλια. Γιατί όταν μιλάμε για κάποια περιθώρια, οροφές ε, και είδους πόρους, πρέπει να ξέρουμε ότι όλα αυτά θα πρέπει να τα επικυρώσουν και τα εθνικά κοινοβούλια. Άρα αυτό το οποίο χρειάζεται είναι πολιτική ηγεσία που θα βοηθήσει την Ευρώπη να υπερπηδήσει αυτή την κρίση και να προετοιμαστεί για την επόμενη φάση. Επομένως, ε, τα τελευταία μου λόγια τα απευθύνω σε όλους, σε όλους μας. Να κάνουμε όλη την απαιτούμενη προσπάθεια για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τη νέα γενιά, για τις επόμενες γενιές για να δείξουμε στους πολίτες των χωρών μας ότι ξέρουμε πώς μπορούμε να ξεπερνάμε κρίσεις και μπορούμε να προετοιμάσουμε την Ευρώπη τον 21ο αιώνα. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιπρόεδρε. Ευχαριστώ. Για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση, η κυρία Υπουργό Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη Ευρωβουλευτέ. Καταρχήν σα ευχαριστώ για τη συζήτηση. Και θα μεταφέρω τις αποφάσεις, τις ε, παρατηρήσει στο Συμβούλιο. Όπω σα είπα, ήδη έχουμε ξεκινήσει το Συμβούλιο το προπαρασκευαστικό έργο βάσει των προτάσεων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δημιουργήσουμε τι προποθέσει για την ε, λήψη απόφαση το συντομότερο δυνατό. Όπω ε, είπα, χθε είχαμε ήδη μία ε, τηλεδιάσκεψη με του Υπουργού Εξωτερικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και εκεί συζητήσαμε κάποια στοιχεία που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ε, για την εφαρμογή των μηχανισμών για να επανεκκινήσει η ευρωπαϊκή οικονομία. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την συνέ... τη συνοχή, τη σύγκληση, την αλληλεγγύη, την ευελιξία και έτσι θα ενισχύσουμε την εσωτερική αγορά, την ανθεκτικότητα και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε μελλοντικέ προκλήσεις. Επίσης θα πρέπει να έχουμε άμεσα διαθέσιμα κονδύλια και σε επαρκή ποσά θα είναι σημαντικό για την αξιοπιστία μας να αντιμετωπίσουμε άμεσα την κρίση. Οι σχετικέ συζητήσει θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρε και εβδομάδε σε όλα τα επίπεδα του Συμβουλίου. Και Ελπίζω να υπάρχει σύγκληση των απόψεων των κρατών μελών, ώστε να έχουμε έγκαιρα συμφωνία, εμπρόθεσμα και για τον επόμενο κοινοτικό προπολογισμό που θα συζητήσει το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο θα χρειαστεί τι κατευθυντήριε γραμμέ από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πριν διαμορφώσει τη θέση του. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εστερνίζεται την ε, ε, δική μα άποψη ότι είναι επίγουσα η ε, έγκριση του προπολογισμού για να καλυφθούν οι ανάγκες και των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών. Γι' αυτό προσβλέπουμε σε συνεχή και καρποφόρο συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να προετοιμάσουμε το έδαφος για ένα φιλόδοξο ε, πιδελταπί που θα στρέφεται στο μέλλον και θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε τρέχουσες αλλά και μελλοντικές προκλήσεις. Ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η συζήτηση. Τα πρακτικά της σημερινή συνεδρίασης ε, θα υποβληθούν για έγκριση στην επόμενη συνεδρίαση. Η συνεδρίαση διακόπτεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.